Good morning, everybody, and most welcome to, to this hearing, this workshop on the protection. Σας καλωσορίζω λοιπόν για την προστασία των ανθρώπων με αναπηρίες. Οργανώθηκε από την Επιτροπή Δικαιωμάτων, όπως επίσης Δικαιωμάτων των Πολιτών να σας ενημερώσω ότι υπάρχει διευμηνία σε όλες τις επίσημες ε, γλώσσες με κάποιες εξαιρέσεις κροατικά, τσεχικά, εσθονικά, φιλανδικά, λιθουανικά, πορτογαλικά και σλοβενικά. Έχουμε επίσης και στην γλώσσα ε, of the fact that this workshop Έχουμε επίσης διαμηνία στη νοηματική αλλά έχουμε και το λεγόμενο velotyping. Όπως είπα είναι ένα τμήμα ενός ετησίου κύκλου εκδηλώσεων ε, στα πλαίσια του ρόλου προστασίας μέσα από την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Αναπηρίες. Όπως ξέρουμε είναι η πρώτη συμφωνία των Ηνωμένων Εθνών που ασχολείται με τέτοια θέματα και είναι η πρώτη επίσης διεθνή συνθήκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα την οποία συνήψε η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μεμονωμένα κράτη-μέλη ταυτόχρονα έτσι ώστε οι πολίτες με αναπηρίες να μπορούν να την χάνουν του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους ισότιμα με όλους τους άλλους. Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με την Επιτροπή Ατομικών Ελευθεριών και τη δική μας Επιτροπή Αναφορών αντιπροσωπεύουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πλαίσια στο πλαίσιο Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Εθνών. Το πλαίσιο αυτό προστατεύει και παρακολουθεί την εφαρμογή της σύμβασης σε θέματα ευρωπαϊκής αρμοδιότητας. Η κυρία Ρώσα Έσταρας Φεραγκούτ αντιπροσωπεύει την Επιτροπή Αναφορών στο πλαίσιο αυτό και σήμερα θα προεδρεύσει του πρώτου τμήματος της συνάντησης αυτής. Δεν έχει φτάσει ακόμα λόγω της κυκλοφορίας της αυξημένης, δεν ξέρω, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε και θα την αντικαταστήσω μέχρι τη στιγμή που θα είναι μαζί μας. Η Επιτροπή μας τα τελευταία χρόνια έχει λάβει πάρα πολύ υψηλούς αριθμούς αναφορών από ανθρώπους με αναπηρίες από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αναφορές αυτές αναφέρονται σε θέματα όπως η προσβασιμότητα, η χρήση της νοηματικής, η επικύρωση της συνθήκης του Μαρακές, η πρόσβαση στην παιδεία, στην εκπαίδευση και η πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Η Επιτροπή αυτή ήταν αρκετά δραστήρια επίσης και για άλλα θέματα που έχουν σχέση με τις αναπηρίες, Υιοθετήσαμε την γνωμοδότησή μας τη σχετική με τη συνθήκη του Μαρακές τον Ιανουάριο του 2017 και την, πράξη, την Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας τον Φεβρουάριο του 2017 τον προηγούμενο μήνα υιοθετήσαμε και μια γνωμοδότηση για τη στρατηγική εφαρμογή γύρω από την αναπηρία στην Ευρώπη μετά από την έκθεση που προετοίμασε και η Επιτροπή Απασχόλησης. Εμείς λοιπόν έχουμε κάνει αρκετά πράγματα νομίζω μέχρι τώρα και πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι. Εδώ έρχεται και είναι ευτυχή στιγμή η διοργανική συμφωνία εφαρμογής της συνθήκης του Μαρακές. Θέλουμε ε, πάντως η συνθήκη αυτή το ταχύτερο δυνατόν να επικυρωθεί από την Ένωση και όλα τα κράτη-μέλη της. Στη σημερινή ε, ομάδα θα ξεκινήσουμε με τη μελέτη την οποία εμείς παραγγείλαμε στα πλαίσια του Τμήματος Μελετών για ε, την ε, εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμού για τους ανθρώπους με αναπηρίες. Ο καθηγητής Έμπερσολντ είναι ένας από τους συγγραφείς της μελέτης, είναι γνωστός κοινωνιολόγος και ερευνητής που έχει δημοσιεύσει πάρα πολλά άρθρα για το θέμα των αναπηριών και του αποκλεισμού των αναπήρων. Αφού τον ακούσουμε θα συνεχίσουμε με δύο πάνελ εμπειρογνωμόνων. Το πρώτο πάνελ είναι το ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο, η σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Συμφωνία των Ηνωμένων Εθνών και το δεύτερο πάνελ νομική ε, και κοινωνική προστασία των ανθρώπων με αναπηρίες. Το πρώτο τμήμα θα το προεδρεύσει η κυρία Ιστάρα Φαραγκούτ, αν τα καταφέρει, η οποία αντιπροσωπεύει την Επιτροπή μας, όπως είπα, στο πλαίσιο συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Εθνών, UNRPD, και στο δίκτυο των αναπηρίων. Και το δεύτερο πάνελ θα είναι πρόεδρος η Μικαέλα Τζουφρίδα. Θα δώσω το λόγο λοιπόν στον καθηγητή Έμπερσολντ για την παρουσίαση της μελέτης. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο και που μου δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσω την ε, δουλειά που έχουμε κάνει για την ε, χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση για ε, μαθητές με αναπηρίες. Καταρχάς, ε, σημαντικό είναι να έχουμε κατά νου ότι χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση δεν ε, έχει διεθνή ορισμό και ένας από τους λόγους είναι ότι η χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση και γενικότερα η εκπαίδευση αποτελεί εθνική αρμοδιότητα. Και η έννοια διαφέρει από χώρα σε χώρα ανάλογα με ε, τον ε, τρόπο που έχει δομηθεί το σύστημα εκπαίδευσης. Δεν υπάρχει λοιπόν διεθνής ορισμός της χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης. Ωστόσο, ε, μια ισχυρή τέτοια εκπαίδευση αποτελεί και σημαντικό πολιτικό στόχο για τα κράτη-μέλη. Και η δουλειά μας δείχνει ότι χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση όχι μόνο αποτελεί προτεραιότητα για τις ε, διάφορες χώρες, αλλά πολλές από αυτές, πολλές χώρες ε, αύξησαν τις δαπάνες τους ε, για την εκπαίδευση αυτή παρά την οικονομική ύφεση. Πολλοί φοβούνται ότι χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση μπορεί να ε, ε, περιοριστεί λόγω των οικονομικών δυσκολιών, αλλά αυτό δεν ισχύει πάντα και μάλιστα πολλές χώρες, πολλές αύξησαν τις δαπάνες. Άλλο σημαντικό θέμα είναι ότι οι χώρες ε, στηρίζονται από διεθνείς οργανισμούς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από την UNESCO για παράδειγμα. από τον ΟΗΕ μέσω της σύμβασης στην οποία μόλις αναφερθήκατε, αλλά και μέσω ε, δραστηριοτήτων όπως είναι η αλληλοδιδαχή ε, και το μοίρασμα, των, ε, τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών. Η χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση σε σχεδόν όλες τις χώρες ε, στόχο έχει να ε, συνδυάσει την ε, καλή απόδοση με την δικαιοσύνη. Αποτελεί τρόπο να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος σε όλες τις χώρες. Η χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση αποτελεί ανταπόκριση σε όλο και πιο πολύπλοκες ε, και επικοινόμορφες ε, κοινωνίες. Και θα πρέπει να θεωρηθεί όχι εμπόδιο, αλλά ως τρόπο να συγκεράσουμε την καλή απόδοση και τη δικαιοσύνη. Η ποικιλότητα αποτελεί ε, θετικό στοιχείο και η χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση συνδέεται με μια νέα προσέγγιση στην εκπαίδευση η οποία ξεφεύγει από, το πρότυπο, από ένα ενιαίο πρότυπο για όλους προς ε, μια ε, εκπαίδευση προσαρμοσμένη στις ανάγκες ε, του καθενός. Η χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση στόχο έχει να αυξήσει τη δυνατότητα του συστήματος να ανταποκριθεί στις ατομικές ανάγκες του κάθε μαθητή. Νομίζω ότι αυτή είναι πολύ σημαντική αλλαγή, διότι οι δυσκολίες των μαθητών δεν συνδέονται με δικά τους χαρακτηριστικά, αλλά με την ανικανότητα των σχολείων να ε, ε, διδάξει μαθητές με διαφορετικά σημεία εκκίνησης. Έτσι λοιπόν εξετάζονται οι ανάγκες του κάθε μαθητή. Και ο κάθε μαθητής υποστηρίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσής του. Οι δυσκολίες των μαθητών συνδέονται και με την ικανότητα του σχολείου να ανταποκριθεί στις ανάγκες του κάθε μαθητή. Τώρα λοιπόν λοιπόν θέλουμε και σχολεία που να υποστηρίζουν τους ασθενέστερους μαθητές αλλά να παρακινώνουν και τους καλύτερους να πετύχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα ώστε να έχει επιτυχία ο κάθε μαθητής ε, ανάλογα με τις ανάγκες του. Μια τέτοια αλλαγή σημαίνει ότι τα σχολεία θα πρέπει να δημιουργήσουν κλίμα εκπαίδευσης ε, χωρίς ε, αποκλεισμούς ε, και να προσαρμόσει το κλίμα στις ανάγκες του κάθε μαθητή. Σημαίνει στην πράξη ότι τα σχολεία θα πρέπει να εξετάσουν το εκπαιδευτικό περιβάλλον, την οργάνωση του σχολείου, την κατάρτιση των καθηγητών ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες του κάθε μαθητή. Η χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση όμως όχι μόνο συνδέεται με την ε, απόδοση και τις ε, ανάγκες των μαθητών ε, αλλά αποτελεί τρόπο να ε, ασκηθεί το δικαίωμα ε, στην εκπαίδευση. Συνδυάζονται εδώ διάφορες διαστάσεις. Η πρόσβαση του μαθητή στο δικαίωμα αυτό σημαίνει ότι η χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση θα πρέπει να παρέχει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης. Αποτελεί δηλαδή τρόπο για εισαγωγή στην κανονική εκπαίδευση. Και με την εκπαίδευση οι άνθρωποι προστατεύονται διότι αυξάνονται οι ευκαιρίες απασχόλησης με την εκπαίδευση, βελτιώνεται η κοινωνική ένταξη, μειώνεται η φτώχεια και προωθείται και η κοινωνική και πολιτική συμμετοχή. Αλλά αυτό δεν αρκεί από μόνο του. Σημαίνει ότι πρέπει να προσφέρουμε και ίσες ευκαιρίες μάθησης στους μαθητές. και έτσι η χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση θα πρέπει να αποτελεί όχι μόνο τρόπο εισαγωγής στη βασική εκπαίδευση, αποτελεί μια διαδικασία στην οποία συμμετέχει ενεργά ο μαθητής και όπου ε, βρίσκεται στο επίκεντρο και ε, η ευημερία του μαθητή. Για παράδειγμα, κάποιες ε, τεχνικές εκπαίδευσης ε, μειώνουν ε, το επίπεδο στρες του μαθητή. Οι αλλαγές αυτές δηλαδή μπορεί να σημαίνουν ουσιαστικά αύξηση των ευκαιριών μάθησης των μαθητών. Οι ίσες ευκαιρίες μάθησης λοιπόν σημαίνουν ότι θα πρέπει να έχουμε συμμετοχή των μαθητών στις πρακτικές διδασκαλίας. Και αυτό όμως μπορεί να μην αρκεί. Πρέπει να παρέχουμε και ίσες ευκαιρίες ε, σχετικά με τα επιτεύγματα των μαθητών. Δηλαδή, η χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση δεν αποτελεί αυτό σκοπό. Αποτελεί τρόπο ώστε το κάθε άτομο να μπορεί να είναι σωστός πολίτης. Θα πρέπει δηλαδή αυτό να θεωρήσουμε ότι αποτελεί αποτέλεσμα της εκπαίδευσης. Εάν συνδυάσουμε λοιπόν ε, τις ε, ίσες ευκαιρίες ε, μάθησης αλλά και ίσες ευκαιρίες επιτυχίας μπορούμε να συνδυάσουμε τα στοιχεία αυτά και έτσι να προστατεύσουμε το κάθε άτομο μέσα από την επιτυχία του στην εκπαίδευση. και να αποφύγουμε την ε, εγκατάλειψη, την πρόορια εγκατάλειψη του, του σχολείου. Όλα αυτά όμως θα πρέπει να συνδέονται και με ίσες ευκαιρίες για τους πολίτες, διότι η χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση αποτελεί παράγοντα κοινωνικής συνοχής. Ε, ευέλικτες πρακτικές διδασκαλίας επιτρέπει στους μαθητές ε, να αποκτήσουν δεξιότητες για ενεργό συμμετοχή. Η χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό τρόπο να προωθήσουμε ε, την ενεργό κοινωνική συμμετοχή και προωθεί επίσης την αποδοχή της διαφορετικότητας. Και πρέπει η χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση να συνδυάζει ακριβώς αυτές τις τέσσερις διαστάσεις. σε ευκαιρίες πρόσβασης, ίσες ευκαιρίες μάθησης, ίσες ευκαιρίες επιτυχίας και σε ευκαιρίες ε, για τους πολίτες. Σε τι βαθμό λοιπόν η χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση επιτρέπει στους μαθητές ε, να είναι ενεργοί πολίτες. If we take the work done Εάν εξετάσουμε την δουλειά του Ευρωπαϊκού Οργανισμού στις διάφορες χώρες, βλέπετε εδώ ότι στις περισσότερες χώρες οι μαθητές ε, για το 80% του χρόνου, οι μαθητές με αναπηρίες, ε, συμμετέχουν στην εκπαίδευση με άτομα χωρίς αναπηρίες. Θέλουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα συγκριτικό πλαίσιο για να αναλύσουμε την κατάσταση. Μέχρι τώρα μια από τις δυσκολίες ήταν ε, ότι δεν ήταν συγκρίσιμα τα δεδομένα των ε, διαφόρων χωρών. Στο πλαίσιο λοιπόν εξετάσαμε τις πρακτικές ε, στις διάφορες χώρες και εντοπίσαμε το ποσοστό των μαθητών ε, με βάση μια ε, επίσημη απόφαση. Μια πολυτομιακή ομάδα ε, ανθρώπων από το σχολείο αλλά και εκτός του σχολείου αξιολογούσαν τον μαθητή και η απόφαση αυτή αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Σε όλες τις χώρες υπάρχουν μαθητές που περνούν από τη διαδικασία αυτή. Εδώ λοιπόν εξετάζουμε τους μαθητές που, για τους οποίους έχει εκδοθεί τέτοια επίσημη απόφαση και που κατά το 80% του χρόνου τους ε, συμμετέχουν σε κανονικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με άτομα χωρίς ε, ε αναπηρίες. Είναι σημαντικό να τονίσουμε αυτήν την τάση η οποία όμως συνδέεται με συγκεκριμένες ε, στρατηγικές διδασκαλίας. Ευέλικτες ε, στρατηγικές διδασκαλίας και η χρηματοδότηση αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα. Η δουλειά μας έχει δείξει ότι η χρηματοδότηση μπορεί είτε να αποτελεί κίνητρο ή εμπόδιο για την ε, χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση. Ο μηχανισμός χρηματοδότησης ε, λοιπόν δείχνει ότι αυτή τη στιγμή οι χώρες που στηρίζουν ε, ε, εκπαίδευση προσαρμοσμένη στο κάθε άτομο χρηματοδοτούν με τρεις τρόπους την εκπαίδευση αυτή. Ε, χρηματοδοτούν ε, τα σχολεία, χρηματοδοτούν τα άτομα και είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι δεν χρειάζεται επίσημη απόφαση για αυτούς τους μαθητές. Και το τρίτο επίπεδο χρηματοδότησης δίδεται σε μαθητές για τους οποίους δυσκολεύεται το σύστημα εκπαίδευσης να ε, παράσχει επαρκή εκπαίδευση και για τους οποίους υπάρχει ε, επίσημη απόφαση. Εδώ λοιπόν ε, βλέπετε τα ποσοστά των μαθητών για τους οποίους υπάρχει επίσημη απόφαση. και σε κάποιε χώρε βλέπουμε ότι το 16% ε, των αυτών έχουν λάβει τέτοια απόφαση ενώ σε άλλε χώρε ε, είναι πολύ χαμηλότερο το ποσοστό. Ε, αυτό σχετίζεται λοιπόν με τον τρόπο χρηματοδότησης προς τους μαθητές αλλά σημαίνει επίσης ότι η δυνατότητα του εκπαιδευτικού συστήματος ε, να αποφεύγει τους αποκλεισμούς διότι όταν αναλύσαμε ε, τα συστήματα. Ε, είδαμε ότι η χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση βασίζεται σε ένα σύστημα με, ε, όπου συμμετέχουν διάφορες ομάδες αλλά και πολλά επίπεδα, δηλαδή τοπικές αρχές, περιφερειακές αρχές, εθνικές αρχές και είναι σαφές ότι τα συστήματα εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς είναι πολύ πιο πολύπλοκα από τα συστήματα γενικής εκπαίδευσης η εφαρμογή και η αποτελεσματικότητα των συστημάτων αυτών εξαρτάται από τα διάφορα συστατικά του συστήματος, η υγεία, η εκπαίδευση, πώς συνδέονται μεταξύ τους λοιπόν οι διάφοροι τομείς. Αυτή η διασύνδεση αποτελεί σημαντικό παράγοντα ώστε ε, να μπορεί να υπάρχει ε, χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση για τους μαθητές και ε, για τις οικογένειές τους και να ενδυναμωθούν αυτές οι ομάδες. Με άλλα λόγια, η εφαρμογή της χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης εξαρτάται από τις συνέργειες που είναι δυνατόν να δημιουργηθούν. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω ότι η χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση βασίζεται σε ένα θεματολόγιο που να προωθεί συστήματα ευέλικτα ε, και μάλιστα σε όλα τα επίπεδα και πρέπει να υπάρχει προληπτική προσέγγιση ώστε να μην υπάρχουν ε, στρατηγικές απόκλησης σε επίπεδο σχολείων. Και τέλος πρέπει να υπάρχει μηχανισμός ε, λογοδοσίας και ελέγχου που να εξετάζει περισσότερο το σύστημα παρά τον ε, κάθε μαθητή. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω. Thank Σας ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά και νομίζω ότι όλοι πλέον είμαστε περήφανοι που είχαμε την ευκαιρία να σας παρακολουθήσουμε σήμερα. Σας ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας και σας διαβεβαιώ ότι σπανίως ε, σε μια επιτροπή εδώ στο Κοινοβούλιο έχουμε ταυτόχρονα δυνατότητες και βελοτάιπινγκ και ε, νοηματικής γλώσσας ε, σε όλη τη διαδικασία. Είμαι πάρα πολύ περήφανη λοιπόν που ανοίγουμε το δρόμο και σε άλλες επιτροπές και ελπίζουμε να ακολουθήσουν. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δουλειά αυτή που κάνετε. Ε, εξαιρετική έκθεσή σας θα έλεγα. Ε, και για τη συμβολή σας σήμερα. Θα ήθελα να επισημάνω δύο πράγματα τα οποία αναφέρετε και νομίζω ότι ε, σημαίνουν πολλά για μας, ε, όχι μόνο ως πολιτικοί ευθύνοντες αλλά και ως άνθρωποι, ότι η ποικιλομορφία, η ανοχή, ε, προωθούν ε, τη συμπόνια και προωθούν και μια καλύτερη κοινωνία. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη από όλους μας ε, με όποια ιδιότητα και αν έχουμε και επίσης πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε και να σας πω ότι μετά τα 50 ορισμένες φορές νιώθω ότι δεν θα πρέπει να αναφερόμαστε σε άτομα με αναπηρία. Όλοι μια αναπηρία έχουμε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο μετά από αυτή την ηλικία. Ε, βρισκόμαστε εδώ σε ένα παγκόσμιο χωριό λοιπόν και πρέπει να επιδεικνύουμε συμπόνια, ε, να δείχνουμε πάθος και να συμπονούμε ο ένας τον άλλον. Ε, θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στους συναδέλφους για ερωτήσεις, σχόλια και κατόπιν να δώσω και πάλι το λόγο σε εσά καθηγητά Εμπερσόλτ. Η Ρώσα. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Γοητεύτηκα από τα όσα μας είπατε. Ήμουν από αυτές οι οποίες προώθησε τη μελέτη για την εκπαίδευση που συμπεριλαμβάνει τους πάντες, ε, διότι θεωρώ ότι είναι από τους βασικούς μοχλούς ε, που ε, βοηθάει και προωθεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και το κλειδί είναι αυτός ακριβώς σε αυτή τη μορφή εκπαίδευσης. Η ερώτηση μου είναι πολύ συγκεκριμένη. Πράγματι, η εκπαίδευση που περιλαμβάνει τους πάντες είναι ένα πολύ σημαντικό μέσο και σε οικονομικό επίπεδο, γιατί ούτως ή άλλως έτσι δημιουργούμε Ευρωπαίους πολίτες, αλλά είναι και σημαντικό για τις αξίες, γιατί ένα παιδί με αναπηρία έχει κίνητρα, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, αλλά οι υπόλοιποι μαθαίνουν αξίες. Και η ερώτησή μου είναι εξής. Γνωρίζετε σε ποιες περιπτώσεις ε, αντιμετωπίζονται, σε ποια κατάσταση βρίσκεται το κράτος μέλος. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ διαφορετική, διότι η αντίληψή μου είναι ότι αυτή η μορφή εκπαίδευση στην Ευρώπη δεν είναι στα επίπεδα που θα πρέπει να βρίσκεται. Η κρίση έχει οδηγεί σε μια οπισθοδρόμηση, διότι αυτή η μορφή εκπαίδευση θέλει και επενδύσει, χρειάζεται ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα σχολεία και δεν είναι το ίδιο να έχουμε ενισχυτική διδασκαλία σε ένα παιδί ε, τυφλό ή σε ένα παιδί ε, με σύνδρομο Down, σε ένα παιδί με δυσλεξία ή σε ε, ένα παιδί με υπερκοινωτικότητα. Ο καθένα χρειάζεται ένα τελείω διαφορετικό δάσκαλο. Και μόνο ε, έτσι μπορεί να γίνει αυτό. Πηγαίνουν παιδιά σε ειδικά εκπαιδευτικά κέντρα όταν δεν υπάρχει δυνατότητα ενισχυτική διδασκαλία στο σχολείο πολλές φορές ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη και αυτό είναι πολύ σύνηθες, δεν είναι η εξαίρεση όταν υπάρχει μια αναπηρία τελικά το παιδί να μην πηγαίνει στο κέντρο της εκπαίδευσης ε, που περιλαμβάνει τους πάντες που προσφέρει και ενισχυτική διδασκαλία αλλά πηγαίνει σε σχολείο ειδική ε, αγωγής. δεν υπάρχουν λοιπόν αρκετές επενδύσεις σε αυτούς τους καθηγητές που μπορούν να προσφέρουν αυτή την ενισχυτική διδασκαλία ο δάσκαλο, είναι ο δάσκαλο όλων των παιδιών, αλλά τα παιδιά με ειδικέ δυσκολίε χρειάζονται και την ενίσχυση αυτή με τον επιπλέον δάσκαλο. Είναι ένα από αυτά τα σοβαρά ζητήματα και ένα άλλο ερώτημα είναι τι πιστεύετε ότι μπορούμε να κάνουμε εμεί ε, μέσω τη Επιτροπής των Αναφορών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να δώσουμε κίνητρα στα κράτη-μέλη Πρόκειται για κάτι το οποίο είναι απολύτω απαραίτητο αν θέλουμε πραγματικά να τηρούμε όλε αυτέ τι αξίε που πρεσβεύουμε. Εγώ πρέπει να σα πω είμαι και αισιόδοξη αλλά και απεσιόδοξη ταυτόχρονα διότι η Επιτροπή μα είναι πάρα πολύ ευαισθητοποιημένη σε αυτά τα θέματα και πιέζουμε πολύ αλλά όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου όταν αναφέρονται στι αξίε, όλο ο κόσμο τι ξέρει απ' έξω και τι απαγγέλει ε, χωρίς πρόβλημα αναφέρεται στα άρθρα που αναφέρονται στι αξίε ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν όμω πρόκειται να ψηφίσουμε όπως προάλλες με την Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας, ε, ε, πραγματικά ε, μας βαραίνει πολύ να ψηφίσουμε ότι πρέπει να γίνει μετατροπή στις μεταφορές για να υπάρχει πρόσβαση σε όλους, πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες, ότι τα ηλεκτρονικά βιβλία πρέπει να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα. εκεί υπήρχε διαίρεση. 300 ψήφοι υπέρ, 300 κατά, γιατί πολλές φορές αντί να λάβει υπόψη τα συμφέροντα των ατόμων, το Κοινοβούλιο όταν ψηφίζει λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα των επιχειρήσεων. Είμαστε πολύ καλοί στη θεωρία, αλλά στην πράξη νομίζω ότι συμβαίνει αυτό που συμβαίνει και στα κράτη-μέλη. Ε, Στι ομιλίε όλοι υπέροχα πράγματα λένε, αλλά μετά στον προπολογισμό και στην υλοποίηση είναι τελείω διαφορετική υπόθεση. Και νομίζω ότι αυτή είναι η κρίση αξιών που βρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω, θα ήθελα να ξέρω πώ αντιλαμβάνετε εσεί το μέλλον. Ε, ακόμα και το Ευρωπαϊκό Σχολείο των Βρυξελών δεν ε, ε περιλαμβάνει τους πάντες και αυτό ε, μπορούν να σας το πούνε όλοι. Τα παιδιά με προβλήματα, αν και είναι λάθος αυτός ο όρος, ένα παιδί με ε, διαφορετικό δεν μπορεί να φοιτήσει σε αυτό το σχολείο τι μοντέλο θέλουμε. Θα έπρεπε να είναι πρότυπο αυτό το σχολείο. Είναι το Ευρωπαϊκό Σχολείο και εγώ έχω γράψει επανειλημμένο στο Ευρωπαϊκό Σχολείο των Βρυξελών. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε πραγματικά το μέλλον και να δημιουργήσουμε πολίτε με αξίε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ θέλω το παιδί μου να έχει αξίε, όχι να ξέρει τόσο πολλά μαθηματικά. Προέχουν οι αξίε και αυτό μπορεί να το δώσει μόνο μια εκπαίδευση που περιλαμβάνει όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για τα σχόλιά σας και για τις ερωτήσεις σας. Πράγματι, αυτή η μορφή εκπαίδευσης στις αρχές έχει μεγάλη υποστήριξη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ε, Ήδη από το Κομένιους συζητούσαμε αυτή την εκπαίδευση που περιλαμβάνει τους πάντες. Αλλά ε, θεωρώ ότι εξελίχθηκαν πολλά πράγματα θετικά ε, τα τελευταία 20 χρόνια και ότι οι χώρες έχουν ξεκινήσει μια πορεία προς μια ε, εκπαίδευση που περιλαμβάνει τους πάντες, διότι αυτή η εκπαίδευση δεν είναι μόνο αναγνωρισμένο δικαίωμα στα πλαίσια της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών, αλλά είναι επίσης και ένα μέσο προκειμένου να συνδυάσουμε απόδοση και ισοτιμία. Και όταν γίνεται ανάλυση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, διαπιστώνουμε ότι ο δρόμο που έχουν διανύσει τα κράτη-μέλη ε, δεν είναι ο ίδιο. δεν έχουν διανύσει την ίδια απόσταση. Κάποιες χώρες έχουν ε, μια λογική που περιλαμβάνει περισσότερο κόσμο από ό,τι οι υπόλοιποι. Αλλά όλοι είναι στην πορεία για την ε, εκπαίδευση αυτή και είναι στην πορεία διότι η εκπαίδευση αυτή εκφύσεως Σήμαινε ότι θέλουμε να προσφέρουμε τη δυνατότητα να πηγαίνουν σχολείο και τα παιδιά με αναπηρία πλέον εδώ ε, ε, και 10 χρόνια ε, εξετάζουμε πώς το εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να είναι αποτελεσματικό για όλους τους μαθητές. Και νομίζω ότι αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική αλλαγή, διότι σημαίνει ότι η έννοια της εκπαίδευσης που περιλαμβάνει τους πάντες, περιλαμβάνει όλους τους μαθητές και όχι μια μειοψηφία μαθητών. Και νομίζω ότι στην ανάλυση που γίνεται ε, εκ των προτέρων για τις ε, πολιτικές οι οποίες εξελίχθηκαν τα τελευταία 20 χρόνια υπάρχει μια πολύ ισχυρή κίνηση υπέρ της εκπαίδευσης που περιλαμβάνει τους πάντες. Πολύ σωστά επισημάνεται βεβαίως, ε, δεν είναι εύκολο να υλοποιηθεί και έχω την εντύπωση δεν είναι εύκολο να υλοποιηθεί διότι δεν λαμβάνουμε ίσως υπόψη τα πράγματα ε, στο βαθμό της περιπλοκότητας που έχουν. Και αυτό είναι και το εθνικό πλαίσιο. Σημαίνει ότι δεν θέλουμε να κάνουμε σύγκριση των πραγμάτων με απλοϊκό τρόπο, αλλά να δούμε και το πόσο σύνθετα είναι. Να παραδεχτούμε ότι σε κάθε χώρα υπάρχει διαφορετική λογική και λαμβάνοντας υπόψη τη συγκεκριμένη λογική της χώρας θα μπορέσουμε να δούμε σε ποιο βαθμό θα μπορέσουν να υπάρξουν οι συνέργειες μεταξύ των χωρών. Και εδώ θεωρώ ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα μπορούν να διαδραματίσουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Επισύοντα την προσοχή σε ε, διάφορες διαστάσεις. Μία εκ των οποίων είναι το γεγονός ότι πρέπει να υπάρχουν και στοιχεία να υπάρχουν στοιχεία τα οποία θα επιτρέπουν να συγκρίνουμε την κατάσταση των ε, μαθητών που χρειάζονται ε, ειδική αγωγή ε, σε σχέση με το σύνολο του πληθυσμού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε με τις χώρες ακριβώς για αυτά τα θέματα της δυνατότητας σύγκρισης. Διότι αντιθήκαμε ότι σε κάποιες χώρες υπάρχουν στοιχεία για τον αριθμό των μαθητών που έχουν πρόσβαση στην ε, συνήθη εκπαίδευση, αλλά ελάχιστες χώρες έχουν στοιχεία για το ποσοστό επιτυχίας των μαθητών που μπορούν να επιτύχουν με αυτή την εκπαίδευση. Ε, και αυτό φυσικά δεν επιτρέπει να δούμε τι πορεία έχει επιτευχθεί, τι πρόοδος έχει επιτευχθεί όσον αφορά τα δικαιώματα αλλά και όσον αφορά τις παιδαγωγικές πρακτικές. Αυτή λοιπόν είναι μια πολύ σημαντική διάσταση. Μια άλλη σημαντική διάσταση θεωρώ ότι είναι το πώς θα επιστήσουμε την προσοχή των χωρών και νομίζω ότι οι χώρες είναι έτοιμες. Υπάρχει διάθεση να προοδεύσουν, να είναι πιο ε, ευαισθητοποιημένες σε θέματα διακυβέρνησης. Διότι όλοι θυμούνται ότι η εκπαίδευση αυτή ε, προϋποθέτει και μεγαλύτερη ευελιξία, μεγαλύτερη αποκέντρωση των εκπαιδευτικών συστημάτων, αλλά η πιο μεγάλη ευελιξία και η μεγαλύτερη αποκέντρωση των εκπαιδευτικών συστημάτων Προϋποθέτει επίσης και άλλες μορφές διακυβέρνησης που θα επιτρέψουν να ε, έχουμε και ένα όραμα για τις εξελίξεις ε, και για τα όσα θα διευκολύνουν αυτές τις πρακτικές. Και θεωρώ ότι και αυτή είναι μια σημαντική διάσταση. Ε, έχει υπάρξει μεγάλη στήριξη, θεωρώ, και η πλειοψηφία των χωρών δαπανούν πολύ περισσότερα για την ε, εκπαίδευση που περιλαμβάνει τους πάντες τη σήμερα ημέρα από ό,τι στο παρελθόν. Ε, έχει αυξηθεί ο προπολογισμό σε πολλές χώρες ε, παρά το γεγονός ότι στη συνέχεια υπήρξαν κάποιες περικοπές στον προπολογισμό. Υπάρχουν λοιπόν επενδύσεις στις χώρες, αλλά αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι οι χώρες δεν τονίζουν και εδώ ίσως θα μπορούσαν να βοηθήσουν τα ευρωπαϊκά όργανα για να ε, δουν ε, πώς μπορούμε να έχουμε κάποια πράγματα τα οποία θα μας επιτρέψουν να ε, κάνουν οι δάσκαλοι αυτό που γνωρίζουν να κάνουν, που πρέπει να κάνουν. Ε, τη στήριξη που πρέπει να δίνεται στα σχολεία, για παράδειγμα, που θα επιτρέπει στα σχολεία να αλλάξουν την οργάνωσή τους. Ε, τη στήριξη στους μαθητές ε, που θα τους επιτρέψει να μπορέσουν να κάνουν αυτό που τους αναλογεί ως μαθητές. Ε, δηλαδή πρέπει να δούμε ε, πώς μπορούμε να περάσουμε από μια λογική που επικεντρώνεται στην ποσότητα που ευνοεί την πρόσβαση στο σχολικό περιβάλλον σε μια ε, διαδικασία που θα ευνοεί την ποιότητα. Και πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, πώς ε, οι παρούσες δομές θα επιτρέψουν στο εκπαιδευτικό σύστημα να προοδεύσει όσον αφορά την εκπαιδευτική του απόδοση. Thank you uh, Um, I Σας ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να θέσω κι εγώ ένα ερώτημα. Εγώ εκτιμώ τη θετική σας αντιμετώπιση. Λέτε ότι τα κράτη-μέλη έχουν επενδύσει πολύ, έχουν ενταχθεί στην οδό της καταπολέμησης του αποκλεισμού. Αλλά τι γίνεται με τα ευρωπαϊκά όργανα Δυστυχώς η κατάσταση στα ευρωπαϊκά σχολεία σχετικά με τα παιδιά με αναπηρίες δεν τα καταφέρνουν καλά και σχετικά με το δικαίωμα των παιδιών στη μαθησιακή διαδικασία και την ένταξή τους στην κοινωνία. Εγώ γνωρίζω πολλά παιδιά σε αυτήν εδώ την πόλη που έχουν εγκαταληφθεί λόγω των αναπηριών τους. Και έχω την εντύπωση ότι είναι πραγματικά ντροπή γιατί τα ευρωπαϊκά όργανα θα έπρεπε να αποτελούν ουσιαστικά τον πρωτοπόρο ε, της αποϊδρυματοποίησης και εμείς έχουμε ε, σαφώς ε, ταξιδέψει σε διάφορες χώρες στα πλαίσια των επισκέψεών μας των διερευνητικών προωθώντας ακριβώς τη μαθησιακή διαδικασία η οποία είναι θα έλεγα ο θεμέλιος λήθος ε, για την ανάπτυξη του παιδιού και το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για τα ευρωπαϊκά σχολεία. Έχετε εξετάσει την υπόθεση των ευρωπαϊκών σχολείων. Όχι μόνο τα έγγραφα, ε, γιατί πολλές φορές υπάρχει μια τεράστια διαφορά ανάμεσα στην πραγματικότητα και στα εξαιρετικά έγγραφα τα οποία μας απασχολούν. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Δεν έχουμε εξετάσει ειδικά τα ευρωπαϊκά σχολεία. Έχουμε συζητήσει το θέμα, αλλά δεν έχουμε κάνει ε, ε, συγκεκριμένες αναλύσεις για τα ευρωπαϊκά όργανα. Έχω την αίσθηση ότι το θέμα των ευρωπαϊκών οργάνων υπογραμμίζει τη μεγάλη σημασία που έχουν, τις που έχουν οι δυνατότητες στήριξης των εκπαιδευτικών αυτών κέντρων. Νομίζω ότι το επίπεδο καταπολέμησης του αποκλεισμού των σχολείων εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο τους επιτρέπουμε να κάνουν κάποια μικρά βήματα. Νομίζω ότι αν η ανάπτυξη αυτή, η ανάπτυξη με τη λογική της συμπερίληψης προχωρήσει σε όλες τις χώρες και προχώρησε σε όλες τις χώρες, αυτό σημαίνει γιατί οι χώρες έχουν δημιουργήσει ένα θεσμικό πλαίσιο που υποστηρίζει τα σχολικά ιδρύματα. Το θέμα το οποίο τίθεται λοιπόν για τα ευρωπαϊκά σχολεία είναι να δούμε τι εξωτερική από το σχολείο στήριξη έχουν έτσι ώστε να μπορέσουν να κάνουν αυτά τα μικρά βήματα προόδου και στον τομέα της προσβασιμότητας και στον τομέα της κατάρτισης. Δεν είναι απόλυτη έννοια η προσβασιμότητα. Η προσβασιμότητα για να υπάρξει, για να συμπεριληφθεί στις οργανωτικές και λειτουργικές λογικές πρέπει να σχεδιαστεί μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Συνεπώς λοιπόν το θέμα αυτό ισχύει για τα σχολεία και ακόμα και τα ευρωπαϊκά σχολεία. Τι είδους στήριξη μπορεί να υπάρξει έτσι ώστε να επιτρέψουμε σε αυτά τα ιδρύματα να κάνουν κάποια μικρά βήματα και να επιδιώξουν την αριστεία ε, συνδυάζοντας τις σχολικές επιδόσεις και την ισότητα ευκαιριών αλλά όλα αυτά προϋποθέτουν, θα έλεγα, ε, υποστήριξη εξωτερική. Νομίζω ότι έχουμε τώρα πια περισσότερα επιχειρήματα για να προωθήσουμε συνολικά και την ιδέα αυτή στα ευρωπαϊκά σχολεία στην πόλη των Βρυξελών. Αυτό είναι κάτι το χρήσιμο αυτά που μας είπατε, έτσι ώστε να είμαστε πιο, θα έλεγα, επίμονοι για τα παιδιά των εκπατρισμένων στις Βρυξέλλες από όλη την Ευρώπη που αντιμετωπίζουν πάρα πολλές δυσκολίες, ιδιαίτερα τα παιδιά τους φυσικά. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε πώς εξελίσσονται τα ευρωπαϊκά σχολεία στις Βρυξέλλες. Σας ευχαριστώ ε, για την παρέμβασή σας. Είμαι ευγνώμων ε, για την ε, παρουσίαση την οποία κάνατε. Το εκτιμούμε δεόντως και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο για την καθοδήγηση του πρώτου πάνελ στην ε, κυρία ιστάρας Φαραγκούτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν το workshop για την προστασία των ανθρώπων με αναπηρίες. Ο στόχος είναι ακριβώς ε, επί τη βάση των αναφορών τις οποίες έχουμε λάβει μέχρι τώρα να μπορέσουμε να δώσουμε κάποιες απαντήσεις. Υπάρχουν πολλές αναφορές ε, για τα θέματα των ανθρώπων με αναπηρία, για τον μη αποκλεισμό από την εκπαίδευση, για την προσβασιμότητα των εκπαιδευτικών δομών, και υπάρχει θέμα επίσης και το θέμα των μεταφορών για τους αναπήρους, υπάρχει το θέμα της χρήσης των νέων τεχνολογιών, υπάρχουν διαφορές στις χώρες σε σχέση με το επίπεδο επιτυχίας ή εφαρμογής αν θέλετε των δυνατοτήτων και των υπηρεσιών που παρέχονται ε, στους αναπήρους. Υπάρχουν διαφορές στις 28 χώρες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 27 από αυτές έχουν επικυρώσει φυσικά ε, την χάρτα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πριν από τον 21ο αιώνα και εκεί προβλέπεται η προστασία των ανθρώπων με αναπηρίες και η χάρτα αυτή αν θέλετε είναι και το πεδίο θα έλεγα αναφοράς μας. Πιστεύουμε ότι η σύμβαση αυτή με την οποία έχουμε δεσμευτεί δεν εφαρμόζεται όπως εμείς θα επιθυμούσαμε και γι' αυτό εμείς προσπαθούμε όπως είπαμε να επιβλέψουμε κάπως τον τρόπο εφαρμογής της σύμβασης σε κάθε κράτος μέλος. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα που θα απασχολήσει το πρώτο πάνελ, του οποίου έχω την τιμή να διευθύνω τις εργασίες τι ακριβώς γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την εφαρμογή της ε, Διεθνούς Συμβάσεως. Η πρώτη ομιλήτρια είναι η Αν Σοφή. Η Αν Σοφή είναι συντονίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τις Αναπηρίες. Είναι ένας ε, ακούραστος εργάτης ε, σε τέτοιου είδους θέματα. Ασχολείται επίσης και με θέματα διακρίσεων εις βάρος των ανθρώπων με αναπηρίες έχει συνεργαστεί με τα Ηνωμένα Έθνη και σίγουρα οι εργασίες της θα διαφωτίσουν την Επιτροπή μας και θα μας δώσουν την δυνατότητα να δούμε αν πράγματι αλλάζουν τα πράγματα και αν ναι προς ποια κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας προς το Ευρωπαϊκό Φόρουμ των Ατόμων με Αναπηρίες. Είμαι η Αν Σοφή από το Ευρωπαϊκό Φόρουμ των Ατόμων με Αναπηρίες και για όσους δεν μας γνωρίζουν, πρόκειται για έναν οργανισμό ευρωπαϊκό για άτομα με αναπηρίες. Εκπροσωπούμε 80.000 άτομα με αναπηρίες και το κάνουμε αυτό κυρίως για να προωθήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τους τελευταίους μήνες σημειώθηκε πρόοδος όσον αφορά την εφαρμογή της σύμβασης. Θέλω όμως να σας μιλήσω και για το τι έχει κάνει ειδικά το Ευρωπαϊκό Φόρουμ πάνω στο θέμα αυτό. Καταρχάς, ε, λοιπόν, δεν βλέπω την παρουσίασή μου στην οθόνη. Δεν πειράζει και πάρα πολύ. Όπως είπε η Ευρωβουλευτής Έστερας, ε, είχαμε την ε, Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία ε, και από την συνάντηση το 2015 οι συστάσεις που προέκυψαν ε, αποτελούν ε, πολύ σημαντικό θεματολόγιο για μας τα τελευταία χρόνια, τους τελευταίους μήνες. Θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο για αυτές τις συστάσεις. Ήδη αρκετοί από τους επιτρόπους έχουν συναντηθεί μαζί μας. Ε, θέλουμε να ε, εφαρμόσουν ε, τα θέματα αυτά στη δουλειά τους. Είχαμε ε, συνάντηση με την ε, Επίτροπο Τίσεν καθώς και τον Επίτροπο Έτιγκερ για να συζητήσουμε ε, την πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ανθρώπινου δυναμικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουμε να υπάρχει περισσότερη υποστήριξη για άτομα τέτοια. Επίσης είχαμε συνάντηση με την Επίτροπο Κρετού διότι στα επόμενα διαρθρωτικά ταμεία θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει αναφορά στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και θέλουμε να βεβαιωθούμε συνεχίσουν να προωθούν τα δικαιώματα αυτά στα κράτη-μέλη. Και τέλο, ε, είχαμε συνάντηση και με τον Επίτροπο Στυλιανίδη. Η τρίτη συνάντηση θα έχουμε μαζί του την επόμενη εβδομάδα, διότι θέλουμε η ε, ανθρωπιστική βοήθεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση επίση ε, να εφαρμόζεται χωρί αποκλεισμού. Θέλουμε λοιπόν να φροντίσουμε και οι πρόσφυγες με αναπηρίες να μην αποκλείονται από την ε, ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και θα ήθελα να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη το 2021 πρέπει να στείλει την επόμενη έκθεση της ε, προς τον ΟΗΕ. Εμείς λοιπόν έχουμε αρχίσει την εκπόνηση της δεύτερης εναλλακτικής έκθεσης που περιλαμβάνει τις απόψεις της κοινωνίας των πολιτών και ατόμων με αναπηρίες σχετικά με την κατάσταση στην Ευρώπη. Κάθε χρόνο οργανώνουμε ακροάσεις ε, της κοινωνίας ε, των πολιτών ε, όπου συμμετέχουν άτομα, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών όπου εξετάζουμε την πρόοδο. λοιπόν είχαμε μια συνάντηση για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα άτομα με αναπηρίες ενώ του χρόνου θα δούμε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως δημόσια διοίκηση. Ε, και λαμβάνουμε αρκετά παράπονα από γονείς και μαθητές των ευρωπαϊκών σχολείων διότι οι μαθητές ε, δεν λαμβάνουν επαρκή υποστήριξη εκεί και γι' αυτό αποστέλλονται και γι' αυτό τους στέλνουν οι γονείς τους σε βελγικά σχολεία και εγώ ως Βελγίδα μπορώ να σας πω ότι και αυτά δεν ε, εφαρμόζουν εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς. Ε, πρόσβαση σε πληροφορίες, σε επικοινωνία από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι θέματα που μας ενδιαφέρουν και ευχαριστούμε την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια για όλη τη δουλειά που έχει κάνει μέχρι τώρα ε, σχετικά με την ευαισθητοποίηση στις ιστοσελίδες Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης και έχουμε και μία έρευνα αυτή τη στιγμή για την ε, ασφάλεια υγείας. Ε, νομίζω ότι σε αυτό θα αναφερθεί η συνάδελφος λίγο αργότερα. Αυτά λοιπόν θα είναι τα θέματα της συνάντησής μας ε, του χρόνου. Και Άλλο σημαντικό θέμα με το οποίο έχουμε ασχοληθεί είναι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα άτομα με αναπηρίες. Νομίζω και ο συνάδελφός μου θα αναφερθεί πιο αναλυτικά στη στρατηγική αυτή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλει έκθεση προόδου ε, με ενδιάμεση αναθεώρηση της στρατηγικής αυτής. Πρόκειται για πολύ χρήσιμο έγγραφο, δίνει μια επισκόπηση της εφαρμογής όλων των ε, διαφορετικών δράσεων και εξετάζει και τις ε, συστάσεις του ΟΗΕ και πόσο έχουμε προχωρήσει όσον αφορά την εφαρμογή αυτών. Επίσης ε, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ ε, έχει συνεργαστεί στενά με το Κοινοβούλιο και την ε, Ευρωβουλευτή Χέλκα Στίβενς. Είχαμε διαλόγους εμπειρογνωμόνων όπου συμμετείχαμε ενεργά και μία από τις βασικές μας ανησυχίες και ένα από τα βασικά μας αιτήματα είναι ότι πρέπει να υπάρξει συνέχεια της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα άτομα με αναπηρίες. Θέλουμε λοιπόν μια στρατηγική που να καλύπτει τη δεκαετία 2020-2030, να καλύπτει όμως περισσότερους από τους 8 ε, κανόνες ε, πολιτικής ε, που καλύπτει αυτή τη στιγμή και θα έχει να κάνει και με την οργάνωση των ανθρώπων με αναπηρίες. Ήθελα να ε, ενημερώσω και σχετικά με την εφαρμογή ε, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία σε εθνικό επίπεδο. Ε, από την Γενέβη έχουν εξεταστεί διάφορες χώρες φέτος Κύπρος, Βοσνία, Ζεγοβίνη, Λουξεμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο, Μαρτενέγρο, Λετωνία, Σλοβενία και η Ισπανία και η Ουγγαρία για δεύτερη φορά και χαιρόμαστε που ε, διάφορα ε, μέλη της οργάνωσής μας συμμετέχουν στην δουλειά αυτή. Απομένουν ε, πολλά να γίνουν όσον αφορά την εφαρμογή αυτών των συστάσεων στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά τουλάχιστον υπάρχουν κατευθυντήρες γραμμές. Άλλο θέμα που παρακολουθούμε στενά Εδώ βλέπετε εικόνες από τα μέλη μας ε, στην ε, Γενέβη που μιλούν ε, στην Επιτροπή για τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία που είναι πολύ καλός τρόπος ευαισθητοποίησης των μελών της Επιτροπής. άλλο θέμα που έχουμε εξετάσει προσεκτικά είναι το Brexit. Το παρακολουθούμε στενά. μαζί με τις ε, οργανώσεις ε, ανθρώπων με αναπηρίες ε, του Ηνωμένου Βασιλείου διότι τα δικαιώματα που έχουν αποκτηθεί μέσω του ευρωπαϊκού δικαίου φοβούμαστε μήπως καταργηθούν πάλι. Εξετάζουμε λοιπόν τα θέματα νομοθεσίας καθώς και το δικαίωμα διαβίωσης εργασίας και σπουδής σε άλλο κράτος μέλος. Εδώ στην οθόνη λοιπόν βλέπετε μία μελέτη όπου εξετάζουμε τις επιπτώσεις του Brexit σε άτομα με αναπηρίες. Παρακολουθούμε στενά τις διαπραγματεύσεις και θέλουμε να φροντίσουμε τα άτομα με αναπηρίες να συμπεριληφθούν στις διαπραγματεύσεις αυτές θέμα που παρακολουθούμε είναι θέματα που σχετίζονται με ε, πρόσφυγες με αναπηρίες. Θα ξανασυναντηθούμε με τον Επίτροπο Στυλιανίδη την επόμενη εβδομάδα για να το συζητήσουμε αυτό από το 2015 και μετά. Πολλά μέλη μας έχουν ε, έρθει και μας έχουν πει ότι στηρίζουν άτομα με αναπηρίες, πρόσφυγες με αναπηρίες που δεν ε, λαμβάνουν επαρκή υποστήριξη. Για παράδειγμα από την Ελλάδα ε, είχαμε την περίπτωση ενός κουφού που δεν ε, μπορούσε να λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες γι' αυτό. Έχουμε δημιουργήσει εντός του Ευρωπαϊκού Φόρουμ μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που θα ασχοληθεί με το θέμα αυτό και που θα βοηθήσει να υπάρξει ευαισθητοποίηση και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε οι πρόσφυγες που ε, διότι πολλοί πρόσφυγες που φτάνουν στα ε, ευρωπαϊκά σύνορα δεν ε, καταγράφονται ως άτομα με αναπηρίες και γι' αυτό δεν λαμβάνουν και την απαραίτητη υποστήριξη ούτε στα κέντρα υποδοχής και σκεφτόμαστε εδώ πέρα θέματα πρόσβασης για παράδειγμα, άτομα ναι, με αναπηρίε μπορεί να μην μπορούν να κάνουν, να μπάνιο, να κάνουν ντους επί ένα μήνα, επειδή δεν είναι σωστά ε, προσαρμοσμένε οι εγκαταστάσει. Ε, Επίσης, άτομα με ε, διανοητική αναπηρία μπορεί να μην λαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες ε, για σχετικά με τα δικαιώματά τους, ε, με την οικογενειακή επανένωση κλπ. Επίσης υπάρχουν πολλοί πρόσφυγες με προβλήματα ψυχικής υγείας λόγω των σκληρών εμπειριών που έχουν περάσει και των κακών συνθήκων στους καταβλισμούς. Έχουμε οργανώσει λοιπόν εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και αλλού ε, διάφορες εκδηλώσεις υψηλού επίπεδου και θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ε, στην Ελλάδα υπάρχει ένα πρόγραμμα σε συνεργασία του ε, οργανισμού, σε συνεργασία με την ε, υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων για τα άτομα με αναπηρίες ε, και ελπίζουμε ότι αυτό θα μπορεί να προωθηθεί και να το μιμηθούν και άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλο θέμα το οποίο με ενδιαφέρει ιδιαίτερα και με το οποίο ασχολούμαι πάρα πολύ είναι τα δικαιώματα γυναικών και κοριτσιών με αναπηρίες, την ισότητα των δύο φύλων. Ε, τους τελευταίους μήνους έχουμε επικεντρωθεί κυρίως σε, θέματα βίασης βάρος ε, γυναικών με αναπηρίες διότι οι γυναίκες με αναπηρίες ε, έχουν τριπλάσιες πιθανότητες να πέσουν θύματα βίας και η επικύρωση της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης είναι κάτι που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Συνεργαζόμαστε στενά με το Ευρωπαϊκό Λόμπι Γυναικών που έχει δημιουργήσει ένα συνασπισμό για ε, ε, την ε, καταπολέμηση της βίας εις βάρος των γυναικών. Και ελπίζουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναλάβει το επόμενο βήμα που θα είναι η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην σύμβαση αυτή. Επίσης, όσον αφορά θέματα στήρωσης και αμβλώσεων γυναικών με αναπηρίες, υπάρχει έχουμε περιπτώσεις ε, αναγκαστικής ε, στήρωσης ε, γυναικών με αναπηρίες Ε, διότι στερούνται των νομικών τους δικαιωμάτων ναι, οι γυναίκες αυτές ε, και αυτό λοιπόν είναι θέμα με το οποίο ασχολούμαστε. Ολοκληρώνουμε σχετική έκθεση που θα παρέχει πληροφορίες και δεδομένα ε, για το θέμα αυτό και θα ζητήσουμε να δοθεί τέλος στην πρακτική αυτή. Και σας προσκαλώ όλους σε ακρόασή μας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 5 Δεκεμβρίου της Ευρωβουλευτής Ραϊπόστ που θα μιλήσει για το που θα ασχοληθεί με το θέμα της στήρωσης κλπ. Άλλο θέμα που θα ήθελα να θίξω είναι η ισότητα και η συμμεταχείριση. Όλοι γνωρίζουμε ότι εδώ και εννέα χρόνια έχει κολλήσει στο Συμβούλιο η σχετική οδηγία. Ε, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ των Ατόμων με Αναπηρία θεωρεί ότι χρειαζόμαστε άλλη στρατηγική λοιπόν και θα δημοσιεύσουμε έκθεση του χρόνου για να, που θα εξετάζει σε τι βαθμό προστατεύονται τα άτομα με αναπηρίες από διακρίσεις σε εθνικό επίπεδο. Θα συγκρίνουμε τα στοιχεία και Ελπίζουμε έτσι να υπάρξει αναβίωση της ε, οριζόντιας οδηγίας για την ίση μεταχείριση. Ε, εδώ βλέπετε την ε, πρώτη, το, το, το πρώτο τεύχος έκθεσης που δημοσιεύσαμε πέρσι σχετικά με την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τώρα λοιπόν θα έχουμε ένα δεύτερο τεύχος και το τελευταίο που θέλω να αναφέρω, το οποίο είμαι βέβαιη ότι θα αναφερθεί πολλές φορές σήμερα, είναι η ευρωπαϊκή πράξη για τα άτομα με αναπηρίες. Η κυρία Εστέρας ανέφερε ότι παρότι είχε υπάρξει πρόοδος σε αρχές Σεπτεμβρίου, ανησυχούμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποκλείονται από την πράξη αυτή και έτσι πολλά άτομα με αναπηρίες δεν θα έχουν πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίε ε, στην σύγχρονη Ευρώπη. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Ιάννη Σοφή. Πράγματι θα είμαστε στις 5 Νοεμβρίου, λέει η Πρόεδρος. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Ρόβερς στην κυρία Ρόβες είχε πολλά χρόνια εμπειρία στις διαδικασίες λήψης απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών οργάνων. Ήταν επίσης και κοινοβουλευτική συνεργάτης κατά τη διάρκεια της έκτης εντολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχετε το λόγο. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω τους οργανητές που προσκάλεσαν και το γραφείο της όμπου της ε, διαμεσολαβήτριας σε αυτήν την συνάντηση σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. Οι εργασίες της διαμεσολαβήτριας ε, καθοδηγούνται θα έλεγα από παράπονα και αναφορές σχετικά με την κακή ε, θα έλεγα διοίκηση στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών οργάνων και των υπηρεσιών. Κάθε πολίτης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή που κατοικεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να καταθέσει ένα τέτοιο, ε, μια τέτοια αναφορά. Το πρόσωπο που καταθέτει την αναφορά δεν χρειάζεται να φύγεται άμεσα προσωπικά ή να έχει νομική υπόσταση. Μπορεί να ξεκινήσει λοιπόν η διαμεσολαβήτρια ε, και δικές της πρωτοβουλίες για ε, συστηματικά προβλήματα στα ευρωπαϊκά όργανα. Στόχος αυτών των πρωτοβολιών είναι να ανταλλάξουμε προτάσεις με τα ευρωπαϊκά όργανα πριν ε, κριθεί απαραίτητο ότι πρέπει να ανοίξει μια επίσημη έρευνα στα πλαίσια επίσης και του πλαισίου παρακολούθησης εφαρμογής του CRPD σε επίπεδο ευρωπαϊκών οργάνων. Έτσι η διαμεσολαβήτρια έχει την ευθύνη να διασφαλίσει ότι η, η διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σέβεται τις παρατηρήσεις των Ηνωμένων Εθνών. Τα θέματα τα σχετικά με την αναπηρία αναφέρονται σε προβλήματα όπως η προσβασιμότητα των κτηρίων, η διαθεσιμότητα υλικού ε, στις ιστοσελίδες, ε, νοηματική ε, διερμηνία σε διάφορα γεγονότα και εκδηλώσεις, όπως επίσης και θέματα κάλυψης των ασφαλιστικών αναγκών στον τομέα της υγείας των παιδιών με αναπηρίες. Έχουμε δύο παραδείγματα εδώ ο τρόπος που αντιμετώπισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την, ε, την ε, διαδικασία επιπαραβάση για την ε, εφαρμογή του CRPD από τις τσεχικές αρχές. Η Επιτροπή είπε ότι το CRPD είναι προγραμματικής φύσεως και θα πρέπει τα κράτη-μέλη ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους να την εφαρμόσουν. Σύμφωνα με τη διαμεσολαβήτρια, οι εξηγήσει ε, ε, ακριβώ παρουσιάζουν ε, τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πότε μπορεί να παρέμβει. Το δεύτερο αφορά τις εικόνες προειδοποίησης στα προϊόντα καπνού. μία από τις εικόνες αυτές δείχνουν κάποιον σε αναπηρική πολυθρόνα, λέγοντας από κάτω ότι το κάπνισμα δημιουργεί προβλήματα αναπηρίας και προβλήματα καρδιαγιακά. Ε, ο αναφέρον διαμαρτύρεται λέγοντας ότι η εικόνα που δίδεται για τις αναπηρίες είναι αρνητική και στιγματίζονται οι ανάπηροι. Ε, η εντολή μας δεν μας επιτρέπει εμείς να ασχοληθούμε με το περιεχόμενο της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, είπε όμως ότι καλό θα είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έρχεται σε επαφή με ομάδες της κοινωνίας των πολιτών πριν επιλέξει τις εικόνες προειδοποίησης. Τώρα θα αναφερθώ σε δύο στρατηγικές έρευνες στον τομέα των αναπηριών. Οι καταληκτικές παρατηρήσεις των Ηνωμένων Εθνών είναι βασικές για μας και για το γραφείο μας. Το 2016 και μετά από τις παρατηρήσεις της Αρμόδιας Επιτροπής και την κατάθεση παραπώνων, ε, η διαμεσολαβήτρια ξεκίνησε μια έρευνα σχετικά με το τι γίνεται με τους αναπήρους στα πλαίσια του κοινού συστήματος κοινωνικής προστασίας του GASIS. Ε, πώς σαν παράδειγμα χαρακτηρίζεται μία ασθένεια ως σοβαρή ασθένεια. Απαιτούνται τέσσερα κριτήρια μεταξύ των οποίων και το κριτήριο ε, μικρότερης αν θέλετε βιωσιμότητας. Νομίζω ότι εδώ ε, ο τρόπος με τον οποίο ε, αντιμετωπίζεται το θέμα των αναπήρων δεν είναι συμβατό με το κοινωνικό πρότυπο το οποίο προωθεί το CRPD. Ιδιαίτερα το κριτήριο της χαμηλότερης βιωσιμότητας δεν είναι το κατάλληλο. Παρ' όλα αυτά ε, οι άνθρωποι αυτοί έχουν τεράστια έξοδα για να καλύψουν τις ανάγκες που διασφαλίζουν την ευημερία των ασθενών τους η διαμεσολαβήτρια ζήτησε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θέσει διαφορετικά κριτήρια για την επιστροφή των εξόδων των ανθρώπων με αναπηρίες. Μετά από μια ανάλυση της ε, απάντησης της Επιτροπής η διαμεσολαβήτρια ζητά συνάντηση με την Επιτροπή. Έγινε μια τέτοια συνάντηση και η έκθεση για τη συνάντηση αυτή δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα μας την προηγούμενη εβδομάδα και συνεχίζεται η έρευνα. Το δεύτερο θέμα του στρατηγικής σημασίας είναι η προσβασιμότητα των ιστοσελίδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ θεωρείται ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχουν ανοιχνευθεί. Το 2016 υιοθετήσαμε και την οδηγία για την προσβασιμότητα ε, των ιστοσελίδων του δημόσιου τομέα. Αυτό δεν ισχύει για τις ιστοσελίδες των ευρωπαϊκών οργάνων, αλλά ζητείτε από, τις, ε, από τα όργανα αυτά να συμμορφωθούν. Και εμείς πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπατε, πρέπει να δείξει το σωστό παράδειγμα. Επίσης προτείνονται χρήσιμα μέτρα τα οποία θα επιτρέψουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αυτές όπως τα θέματα παρακολούθησης, εποπτείας, όπως επίσης και τα θέματα μιας, τα σχετικά με μια δήλωση προσβασιμότητας με πληροφορίες για τους χρήστες. Ξεκινήσαμε τον Ιούλιο του 2017 και μια στρατηγική έρευνα για την προσβασιμότητα των ιστοσελίδων αυτών λοιπόν. Η διαμεσολαβήτρια έστειλε μια επιστολή στον πρόεδρο Γιούνκερ και έθεσε θέματα όπως η αξιολόγηση της προσβασιμότητας των ιστοσελίδων, η παροχή πληροφοριών σε νοηματική γλώσσα, η εκπαίδευση των μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η προσβασιμότητα των εσωτερικών δικτύων, όπως επίσης και το θέμα της δήλωσης προσβασιμότητας. Όλα αυτά είναι υπό εξέταση. Η δημοσίευση της, Επιτροπής, της απάντησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναμένεται σύντομα. Εδώ και αρκετό καιρό έχουμε προσπαθήσει να καταστήσουμε και τη δική μας ιστοσελίδα πιο προσβάσιμη και φιλική στο χρήστη. Ε, εξηγούμε τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε, όπως επίσης και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να καταθέσει κανείς ένα παράπονο ή μία διαμαρτυρία. Ε, επίσης διασφαλίσαμε και την συμβατότητα της ιστοσελίδας μας με το WCAG 2.0 ε, ακριβώς και πήραμε ένα βαθμό συμμόρφωσης 2α. Ε, ε, ταυτόχρονα προσπαθούμε να ε, εκπαιδεύσουμε το προσωπικό μας σε σχέση με την λειτουργία των ιστοσελίδων αυτών. Από τον Ιούλιο μπορείτε να βρείτε μια νέα σελίδα με ενημερώσεις για τις δυνατότητες προσβασιμότητας. Η διαμεσολαβήτρια επανειλημμένα λέγει ότι απαιτείται να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες δράσεις, να μην μείνουμε σε δηλώσεις χωρίς περιεχόμενο για την καθημερινότητα των ανθρώπων με αναπηρίες. Θα συνεχίσει να παίζει λοιπόν συγκεκριμένο ρόλο σε σχέση με την εφαρμογή του CRPD σε κοινοτικό επίπεδο. Και πέρα από τις παρατηρήσεις των Ηνωμένων Εθνών, θα ήθελα να πω ότι είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι όταν ανταλλάσσουμε ε, εμπειρίες όπως σήμερα γιατί αυτό θα βοηθήσει τους πολίτες. Ευχαριστώ πολύ. Θα περιμένουμε βεβαίως και τις απαντήσεις ε, σε όλες αυτά ε, στις ερωτήσεις μέσω των όσων κάνει ε, ο Ευρωπαίος ε, Διαμεσολαβητής. Να δώσουμε τώρα στη, ο λόγο στην Ημακουλάδα Πλασένθια. Είναι μεγάλη εμπειρογνώμονας επί των θεμάτων και είναι και ε, σύμβουλος στην Επιτροπή για θέματα αναπηρίας. Είναι ε, επικεφαλής του τμήματος ε, ατόμων με αναπηρία στο ε, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως γνωρίζετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν ιδιαίτερα φιλόδοξη, πολύ περισσότερο από το Κοινοβούλιο στην Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας και η ίδια ήταν αυτή η οποία πίεσε τρόπον την άπρος αυτή την κατεύθυνση. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω λοιπόν εξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών με την άδεια της Πρόεδρου για την εξαιρετική δουλειά που κάνεις προς όφελος του συνόλου και είναι και υπεύθυνη της ομάδας ε, εργασίας για την κατάρτιση αυτής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για την προσβασιμότητα. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα λοιπόν που είστε εδώ σε αυτό το πάνελ και σας ακούμε. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς για τα πολύ καλά σας λόγια. Και σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση για να μπορέσω να μοιραστώ μαζί σας ε, όλα όσα κάνουμε για την πρόοδο για την εφαρμογή της ε, Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Όπως γνωρίζετε, Τα όσα κάνουμε για την εφαρμογή της ε, σύμβασης ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πλαισιώνονται στα ε, πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Αναπηρία και η οποία ξεκίνησε το 2010 και θα λήξει το 2020. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιτευθούν οι στόχοι της σύμβασης και αυτό συνάδει και με τους στόχους ε, της ενδυνάμωσης των ατόμων με αναπηρία για να μπορούν να απολαμβάνουν πλήρως ε, τα δικαιώματά τους και να υπάρχει και μια Ευρώπη ε, χωρίς φραγμούς. Αυτό είναι αυτό το οποίο προσπαθήσαμε να κάνουμε για την προσβασιμότητα τα τελευταία χρόνια και θα συνεχίσουμε να διαμορφώνουμε και το χαρακτήρα για να υπάρχουν κατάλληλες προϋποθέσεις ε, πρόσβασης στα δικαιώματα. Έχουμε συγκεκριμένου τομείς εργασίας, ε, στους οποίους ε, παρουσιάσαμε και μια γενική εικόνα των βασικών επιτευγμάτων μέχρι το 2017, το Φεβρουάριο του 2017, όπου και δημοσιεύθηκε μια έκθεση πρόοδου. Σε αυτή την έκθεση πρόοδου είχαμε δύο βασικούς στόχους. Πρώτον, να υπάρξει μια εικόνα των όσων κάναμε εμείς τα πρώτα χρόνια και δεύτερον, να βρούμε τις κατάλληλες απαντήσεις και να δείξουμε πώς ε, απαντάμε στις συστάσεις που δόθηκε από την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να γίνει αυτό, η έκθεση είχε τα βασικά στοιχεία και θα σας δώσω και μερικά παραδείγματα εντός ολίγου σε μια προσπάθεια να σας δείξω και τι ακριβώς ε, ε, αναβαθμίσαμε φέτος και περιλαμβάνει και μια σειρά από ε, σημαντικά παραρτήματα. Καταρχάς έχουμε μια εικόνα της δημόσιας διαβούλευσης και φέτος η δέσμευσή μας ε, και η επικοινωνία μας με άτομα με αναπηρία, οργανώσεις που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρία και γενικώ ε, ε, ε, οποιονδήποτε εργάζεται με άτομα με αναπηρία και φυσικά και κράτη-μέλη και δημόσιες αρχές είναι πάρα πολύ σημαντική για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έγινε η δημόσια διαβούλευση, είχαμε πάνω από 1.500 απαντήσεις και οι ανησυχίες που εκφράστηκαν ήταν καταρχάς ε, έλλειψη πρόσβασης σε θέσεις εργασίας και πρόβλημα με τις μεταφορές. Οι γνώση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, ευαισθητοποίηση για την ε, γνώση των δικαιωμάτων, αυτά ήταν ε, πολύ σημαντικά στοιχεία που μας απασχόλησαν κατά την εφαρμογή της σύμβασης. Προχωρούμε με διάλογο με την κοινωνία των πολιτών. Φέτος έγιναν αρκετές συναντήσεις με οργανώσεις της κοινωνία των πολιτών για να παρακολουθήσουμε αρκετά από αυτά τα θέματα. Το δεύτερο παράρτημα είναι μια περιγραφή όλων των δράσεων. Έχουμε πάνω από 100 δράσεις οι οποίες συνοδεύουν αυτή τη στρατηγική και αναφέρεται τι κάναμε και τι εκκρεμεί. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι φέτος ε, ε, υπήρξε μια συνέχεια σε κάποιες από αυτές τις δράσεις. Να πω επίσης ότι το παράρτημα 3 περιλαμβάνει τις συγκεκριμένες συστάσεις, να υπάρχει συγκεκριμένη απάντηση δηλαδή σε κάθε μία από τις συστάσεις που λάβαμε και τέλος ε, είδαμε και τι κάνουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το επισημάνομαι, είναι ένα τομέας στον οποίο παρακολουθούμε ε, ο εκπρόσωπος της ε, διαμεσολαβήτριας αναφέρθηκε στις ιστοσελίδες, με την προσβασιμότητα των ιστοσελίδων, υπάρξει παρακολούθηση, υπήρχαν και εκπαιδευτικά προγράμματα, μαθήματα κατάρτισης ε, και κάθε φορά που δημοσιεύεται μια νέα ιστοσελίδα προσπαθούμε να δούμε και να ελέγξουμε την προσβασιμότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι εξετάζουμε το θέμα αυτό ε, και παρά το γεγονός ότι το ανέφερε και ο εκπρόσωπος της και αυτό αφορά όχι μόνο τους ε, υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά όλους τους αξιωματούχους ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα τα θεσμικά όργανα και είναι πάρα πολύ σημαντικό και το λαμβάνουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη. Τέλος, να αναφερθώ στο τελευταίο παράρτημα, που περιλαμβάνει τις δράσεις εξορθολογισμού που ε, είχαμε όταν θέλουμε να εφαρμόσουμε τη σύμβαση και όταν αναφέρω με στις δράσεις αυτές αφορούν και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και εσά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν εγκρίνετε νομοθετικές πράξεις. Το 2010 η δήλωση αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιελάμβανε περίπου 45 με 46 νομικές πράξεις ε, ε, που ε, προσπαθούσαν να συμπεριβλάβουν και την αναπηρία. Τώρα έχουμε πλέον 230 νομικές πράξεις που περιλαμβάνουν αναφορές και στην αναπηρία και θα σας δώσω και κάποια παραδείγματα για κάποιες πρόσφατες εξελίξεις οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα. Εξετάζοντας τα βασικά στοιχεία του εγγράφου, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι ακόμα έχουμε πάρα πολλές εκκρεμότητες Δεν δουλεύει και το μηχανηματάκι, τώρα δουλεύει. Uh, yes. Okay. Well, that one. Okay. Uh, ποτέ δεν δουλεύουν αυτά τα μαραφέτια, τα καταφέραν. Τώρα λοιπόν καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι στόχοι της στρατηγικής εξακολουθούν να μας αφορούν και για την επόμενη πενταετία, γι' αυτό ακριβώς και προσπαθήσαμε να ε, τους προωθήσουμε και το 2017. Η προσβασιμότητα είναι ένας από τους τομείς ε, στον οποίο αφιερώνουμε τις περισσότερες προσπάθειές μου. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Πράξη προσβασιμότητα και προσπαθούμε να διατηρήσουμε το καλό επίπεδο που θεωρούμε ότι περιλάμβανε η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα βασικά στοιχεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει πρόσβαση για τα άτομα με αναπηρία, αυτή που χρειάζεται, αλλά να αναφερθώ και στα όσα γίνονται σε επίπεδο υλοποίηση. Παραδείγματο χάρη στην οδηγία για την προσβασιμότητα στο διαδίκτυο πριν τεθεί σε ισχύ. Υπάρχουν κάποιε κατευθυντήριε γραμμέ που πρέπει να προωθήσουμε και να υπάρχουν και εκτελεστικά μέτρα. Δεν ε, θα σα αναφέρω μία προς μία τις πρωτοβουλίες, αλλά θα αναφέρω κάποιες εξ αυτών. τα πιο βασικά για τον κάθε τομέα. Στον τομέα της συμμετοχής, για παράδειγμα, προχωρούμε καλά με την πρωτοβουλία για να έχουμε έναν Ευρωπαίο φύλακα αναπηρίας. Είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, διότι πρέπει να την προωθήσουμε μαζί με τα κράτη-μέλη. Αυτά έχουν την αρμοδιότητα, αλλά συνεργαζόμαστε για να υπάρχει μια κάρτα, ευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας, για να μπορεί κάποιο να απολαμβάνει συγκεκριμένα δικαιώματα ε, και όσον αφορά τον ορισμό της αναπηρίας ε, βοηθούμε τα κράτη-μέλη για να διοργανώσουν συγκεκριμένα εργαστήρια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα και η σύμβαση ακόμα δεν έχει διευκρινίσει πώς μπορούμε να κάνουμε καλή αξιολόγηση η οποία θα αντανακλά και την πρόσβαση ε, και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι κάτι το οποίο είναι πάντα προϋπόθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Συνεργαζόμαστε λοιπόν με τα κράτη-μέλη ε, τα οποία αυτή τη στιγμή ε, κάνουν τη σχετική εργασία για το πώς μπορούν να το υλοποιήσουν. Για να γίνει αυτό Έχουμε ένα δίκτυο εμπειρογνωμόνων, έχουμε συλλέξει πληροφορίες, συνεχίζουμε να συλλέγουμε πληροφορίες από τα κράτη-μέλη. Να σταθώ επίσης και στον τομέα της ε, κοινωνικής προστασίας, ε, το πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων. Το έχω βάλει στα θέματα της κοινωνικής προστασίας γιατί το θέμα της αναπηρίας ε, συγγενεύει με όλα αυτά. Ε, μαζί με τους εμπειρογνώμονες μας φέτος προσπαθούμε να συλλέξουμε στοιχεία για να έχουμε κάποιες συστάσεις για το πώς μπορούμε να εξορθολογήσουμε καλύτερα και να συμπεριλάβουμε ε, θέματα αναπηρίας σε όλα αυτά ε, των πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων και ε, να δούμε όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την αναπηρία. Για να τονίσω και μία πολύ σημαντική εξέλιξη στην πρωτοβουλία που συνόδευε τον πυλόν αυτό, η ισορροπία εργασιακού και οικογενειακού βίου, ε, για πρώτη φορά υπήρχε σύσταση όχι μόνο να προσέξουμε γονείς που έχουν άτομα με αναπηρία ή που είναι ε, υπεύθυνοι για τη φροντίδα ατόμων με αναπηρία αναφέρονται και σε γονείς με αναπηρία που ε, πολύ συχνά ε, χρειάζονται και κατάλληλα μέτρα και μπορούν να φροντίσουν τις ανάγκες τους. Και θα ήθελα να κλείσω με μια αναφορά στα όσα γίνονται για την εξωτερική δράση. Συνεχίζουμε με ένα πρόγραμμα για την ανάπτυξη δικτών που συνδέουν, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, τη σύμβαση με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Να υπάρχουν δείκτες για τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης που αντανακλούν και τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στη σύμβαση. Ε, και αυτό αποτελεί ένα ακόμα παράδειγμα. Νομίζω δεν έχουμε και πολύ χρόνο και θα ήθελα να πω ότι εξακολουθούμε με τις πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης, το ετήσιο φόρουμ για την ερμογή της σύμβασης ε, συζητά με τη συμμετοχή όλων των εθνικών ε, σημείων εστίασης, τους μηχανισμούς συντονισμού και ανεξάρτητους μηχανισμούς ε, και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ζητήσουμε σημαντικά στοιχεία όπως πρόσφυγες με αναπηρία, πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα άρθρα της σύμβασης που αφορούν το θέμα αυτό και επίσης και την αξιολόγηση της αναπηρίας. Ολοκληρώνοντας να πω απλώς ότι θα συνεχίσουμε να προωθούμε την εφαρμογή της σύμβασης ε, στα πλαίσια της στρατηγικής και θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τις συστάσεις ως ε, ε, πηξίδα, αλλά αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι επειδή η στρατηγική περιλαμβάνει συγκεκριμένες δεσμεύσεις ε, ε, και νέες πρωτοβουλίες που περιλαμβάνουν θέματα συμπερίληψης και των, ε, της αναπηρίας. Για παράδειγμα, στην οδηγία και τη σχετική νομοθεσία για τα δικαιώματα των επιβατών των σιδηροδρόμων προσπαθήσαμε να συμπεριλάβουμε και την προσβασιμότητα. Συζητούμε επίσης και με την κοινωνία των πολιτών, αλλά για του χρόνου θα επικεντρωθούμε επίσης και σε μία περίοδο προβληματισμού για να προετοιμαστούμε, να αξιολογήσουμε και να έχουμε και μία πολύ καλή εικόνα των αποτελεσμάτων της στρατηγικής ώστε να ε, προετοιμάσουμε τα επόμενα βήματα και μετά το 2020 και να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες ε, για να ξεκινήσουμε να προετοιμάζουμε την περιοδική έκθεση πρόοδου που ε, αναμένεται το 2021. Και εδώ θα ήθελα να τονίσω ε, και να ευχαριστήσω για τα όσα κάνετε εσείς εδώ στο Κοινοβούλιο ε, για την έκθεση που αναφέρθηκε και προηγουμένως για την πρόοδο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Αναπήρεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και ε, σε περίπτωση που υπάρχουν ερωτήσεις είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Μακουλάδα. Με αυτό λοιπόν ολοκληρώνεται το πρώτο πάνελ και με την άδεια της Προέδρου θα περάσουμε στο επόμενο πάνελ, το οποίο θα συντονίσει η Μικαέλα Τζουφρίντα. Ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Χαίρομαι που ως αντιπρόεδρος της Ομάδας για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ως μέλος της Επιτροπής προεδρεύω σε αυτό το πάνελ. Η Επιτροπή Αναφορών είναι σημείο αναφοράς και εμείς ως άμεσοι συνομιλητές με τα άτομα με αναπηρία και με τις οργανώσεις που τα εκπροσωπούν είμαστε σε προνομιούχα θέση διότι είναι πάμπολοι οι πολίτες που απευθύνονται σε αυτή την Επιτροπή. Ο σεβασμός της αξιοπρέπειας, της αυτονομίας, της ανεξαρτησίας των ατόμων, των ίσων ευκαιριών, ε, της έλλειψης διακρίσεων είναι ε, προϋποθέσεις τις οποίες σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να λησμονούμε. Τα άτομα με αναπηρία θα πρέπει να χαίρουν όλων των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Πραγματικά λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους που είναι εδώ παρέντε σήμερα και θα συμμετέχουν σε αυτό το και εκτίμησα ιδιαίτερα και όλα όσα άκουσα μέχρι τώρα, τις παρουσιάσεις που ακούσαμε. Έχουμε εκπροσώπους των οργανώσεων που ε, συνεργάζονται συνεχώς ε, σε πολύ αισθανή επαφή με τα άτομα με αναπηρία και οι μαρτυρίες τους, η συμβολή τους και το γεγονός ότι μπορεί να υπάρξει μια αγώνιμη αντιπαράθεση είναι πάρα πολύ σημαντικά για τη δουλειά μα για το έργο των θεσμικών οργάνων. Στο Κοινοβούλιο το Σεπτέμβριο σε πρώτη ανάγνωση και από πολύ μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε η Ευρωπαϊκή Πράξη για την Προσβασιμότητα των Αναπήρων και όπω ξέρετε περιλαμβάνονται και κάποιε συγκεκριμένε προποθέσει προσβασιμότητα για αγαθά και υπηρεσίε που κυκλοφορούν στην ενιαία αγορά. Πρόκειται για την αρχή μια πορεία την οποία θέλουμε και πρέπει να προωθήσουμε και χάρη στην αντιπαράθεση και την ανταλλαγή πληροφοριών με τις οργανώσεις των εκπροσώπων των ατόμων αυτών. Οι πολιτικέ για την αναπηρία που θέλουν να έχουν μια πιο καλή βοήθεια, την αναγνώριση του ρόλου των ατόμων που προσφέρουν φροντίδα ε, και φυσικά όλα αυτά περιλαμβάνονται στου στόχου μα και είμαι βέβαιη ότι ε, εργαζόμενοι ε, όπως πάντα με μεγάλη ε, ένταση θα καταφέρουμε να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους. Σε αυτή τη δεύτερη συνεδρία θα ακούσουμε άτομα από οργανώσεις που εργάζονται σε πολύ στενή επαφή με άτομα με αναπηρία. Έχουμε εκπροσώπους του Inclusion Europe, του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Ανεξάρτητη Διαβίωση και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ατόμων που παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρία. Ε, θα ήθελα εδώ να αναφέρω λοιπόν τον κύριο Ζακινό, ο οποίος είναι αρμόδιος για τις πολιτικές ε, στο Inclusion Europe, τη Ζάρα το Ζάρα Τόντ που είναι διευθυντής του ΕΜΙΛ που είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για μια αυτόνομη ζωή και τον Τόμας Μπινιάλ ο οποίος είναι υπεύθυνο πολιτικής για την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Παρόχων Υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρία. Θα ήθελα να ζητήσω ευγενικά από τους ομιλητές να σεβαστούν το χρόνο αγόρευσης που τους έχει ε, διατεθεί, 10 λεπτά υπενθυμίζω και μετά θα περάσουμε σε ένα ε, γύρο ερωτήσεων και απαντήσεων. Παρακαλώ κύριε Ζακινό, έχετε το λόγο. Thank you, uh, Mrs. Uh, Griffrida. Um, Ευχαριστώ κυρία Τζοφρίδα. This invitation today. Um, what is love? in a court to decide if it... Τι είναι η αγάπη γιατί αυτοί που ψηφίζουν παίζουν ρόλο για σας, έχουν σημασία για σας. Γιατί τέθηκε και το ερώτημα σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν διανοητικές δυσκολίες για το αν είναι ικανοί και σε ποιο βαθμό είναι ικανοί να επιλέγουν στις εκλογές. Γι' αυτό λοιπόν η προτεραιότητα σε εμά είναι η στέρηση της νομικής προσωπικότητας και σε ποιο βαθμό αυτό επηρεάζει την απώλεια ελέγχου της καθημερινότητας. Εξ ονόματος των 7 εκατομμυρίων ανθρώπων με διανοητική αναπηρία μαζί με τις οργανώσεις των γονέων 71 πρακτικές από 31 χώρες είναι στην ουσία αυτό που καταγγέλουμε τα στερεότυπα που στερούν την δυνατότητα από τους αναπήρους να ε, γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά τους στην οικογενειακή ζωή, στην ε, αισθηματική του ζωή, στην κατοικία, όπως είπε και η Ανσοφή προηγουμένως σε άλλους τομείς. Δεύτερο θέμα είναι η ιδρυματοποίηση. Απομονώνονται μέσω της ιδρυματοποίησης ένα εκατομμύριο Ευρωπαίοι το χρόνο. Ιδιαίτερα αυτοί που έχουν διανοητικού τύπου θέματα. Και στην ουσία τα παιδιά που πηγαίνουν στα ιδρύματα στερούνται την οικογένειά τους και στερούνται την οικογένεια, την δυνατότητα να, κάνουν, να έχουν κανονική οικογενειακή ζωή και σχολική ζωή του στερείται το δικαίωμα της ιδιωτικότητας, το δικαίωμα ίδρυσης μιας οικογένειας και τέλος υπάρχει το θέμα της έλλειψης κατανοητών ε, προσπαθειών ενημέρωσης που επηρεάζει τους ανθρώπους αυτούς και τους απαγορεύει να συμμετέχουν σε κοινωνικές διαδικασίες και να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες. Όπως είπε και η προηγούμενη εμιλήτρια, σαν παράδειγμα η έλλειψη γνώσεων των ανθρώπων με αναπηρίες για τα δικαιώματά τους είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να καλυφθεί από την κοινωνία των πολιτών. Και αυτά καλύπτονται και από τις οδηγίες που έχετε σήμερα. Σαν παράδειγμα το θέμα που θα συζητήσετε σήμερα για την Αυστρία ε, άπτεται του πώς οι διαθέσιμες πληροφορίες επηρεάζουν την καθημερινότητα. Η αναφορά από την Ιρλανδία δείχνει ότι οι οδηγίες για τη γεωργική δραστηριότητα δεν είναι κατανοητές ενώ απαιτείται από όλους, ενώ απαιτείται από όλους να γίνονται σεβαστές. ιδιαίτερα αυτοί οι οποίοι έχουν στην οικογένειά τους ε, και ε, παιδιά και γυναίκες με διανοητικές δυσκολίες που υφίστανται διπλά και τριπλά επίπεδα διάκρισης. Θα πρέπει λοιπόν να βοηθηθούν οι άνθρωποι αυτοί να μπορέσουν να αυτοκαθορίσουν την εξέλιξη της ζωής τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το 2000 την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα προώθησης των προσωπικών συμφερόντων ανθρώπων οι οποίοι έχουν αναπηρίες αλλά θέλουν να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Πολλοί από αυτούς θέλουν να είναι και είναι καθηγητές, δάσκαλοι, παροχή υπηρεσιών και πανεπιστημιακοί και θέλουν να βοηθήσουν όλους τους ανθρώπους με τέτοιου είδους αναπηρίες. Σαν παράδειγμα τα μέλη μας στην Ουγγαρία συνεργάζονται με την αστυνομία έτσι ώστε να υπάρχει σωστή υποδοχή των ανθρώπων με αναπηρίες που υφίστανται βία ή επιθέσεις. Και υπάρχει επίσης και υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο άρθρο 3 της οδηγίας του 2010 για το δικαίωμα στην κατανόηση των διαδικασιών και το δικαίωμα στην έκφραση στη συμμετοχή τους στις διαδικασίες. Να συμμετέχουν λοιπόν στις αποφάσεις οι οποίες τους αφορούν πολλά από τα προγράμματα και τις εκδηλώσεις που οργανώνουμε μέσω των λεγόμενων self-advocates έχουν σαν στόχο να βοηθήσουν Έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο λέγεται Top-Sighted, το οποίο ε, λειτουργεί με τη λογική ε, του μέντορα. Είναι οι μέντορες οι οποίες ε, βοηθούν τους ανθρώπους αυτούς να ελέγξουν τη ζωή τους και να γίνουν δραστήριοι πολίτες. Γι' αυτό λοιπόν έτσι μπορούμε να βοηθήσουμε τους αναπήρους. Προωθούμε επίσης και την ευρύτατη χρήση ε, οδηγιών και πληροφοριών με κατανοητή, εύκολα κατανοητή διατύπωση και μορφή. Έτσι θα επιτρέψουν στους ανθρώπους αυτούς να συμμετέχουν περισσότερο σε σχέση με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για ε, τις μορφές easy to read, για μορφές εύκολης αναγνωσιμότητας ε, και αυτό ε, αφορά επίσης και στις προβλέψεις ε, της πράξης για την προσβασιμότητα. Και επίσης ε, πρέπει να προσπαθούμε να βρούμε και τρόπους ενημέρωσης αυτών που έχουν διανοητικές, διανοητικά θέματα να είναι ενημερωμένοι και να γνωρίζουν τα πράγματα που τους αφορούν και θα πρέπει να βοηθήσουμε και αυτούς οι οποίοι ασχολούνται στα πλαίσια του προγράμματος Self-Advocate έτσι ώστε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Σαν παράδειγμα συναντήθηκαν εκπρόσωποι αυτής της οργάνωσης με εννέα ευρωβουλευτές για να μιλήσουν για την βία εις βάρος των γυναικών στα ιδρύματα ψυχιατρικά. Ε, όλα αυτά λοιπόν οι άπτονται και τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών που έχει επικυρωθεί και πρέπει να εφαρμοστεί σωστά σε όλες τις χώρες. Είναι θέμα όπως βλέπω το οποίο συζητιέται έντονα στα πλαίσια του καθορισμού μιας νέας στρατηγικής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι πολύ πιο φιλόδοξη για την προώθηση των αξιών του CRPD των Ηνωμένων Εθνών παράδειγμα είναι νέοι στόχοι για το κλείσιμο των περισσότερων ιδρυμάτων ε, για να ασχοληθούμε με τα αρνητικά σημεία της στέρησης της νομικής προσωπικότητας και τις συνέπειες που έχει κάτι τέτοιο. Θα πρέπει οι πρακτικές αυτές να είναι παράδειγμα για όλα τα κράτη-μέλη στα πλαίσια της υποχρέωσης εφαρμογής της σύμβασης. Σαν παράδειγμα, οι ιστοσελίδες θα πρέπει να γίνουν της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαδραστικές από την πρώτη μέχρι την τελευταία σελίδα και σε επίπεδο δημόσιας διαβούλευσης και σε επίπεδο σύνταξης προτάσεων και σε επίπεδο γενικότερης παρέμβασης. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια θέματα με τη διανοητική βέβαια αναπηρία Κάποιες από τις ανάγκες τους έχουν αρχίσει να καλύπτονται και αυτό είναι ένα καλό μήνυμα. Επίσης οι πληροφορίες οι οποίες δίδονται στους Ευρωπαίους πολίτες και οι προσκλήσεις προς τους Ευρωπαίους πολίτες θα πρέπει να είναι προσβάσιμες σε όλες τις φάσεις διατύπωσής του. Αυτά στα 10 λεπτά δεν μπορώ να πω περισσότερα. Γι' αυτό τελειώνοντας θα σας θέσω ένα ερώτημα, όχι σαν δικαστής αλλά σαν πολίτης που ανησυχεί. Τι θα κάνετε για να περάσουμε πια σε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Ευχαριστώ κύριε Ζακινό, σας ευχαριστώ ε, για την παρουσίασή σας, σεβαστήκατε το χρόνο σας. Θα δώσω τώρα τον λόγο στην Σαρατόντο για 10 λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω στην Επιτροπή σας. Είμαστε μία οργάνωση που εργάζεται στο σύνολο της Ευρώπης ε, για να προωθήσουμε και να υπερασπιστούμε ε, τα δικαιώματα των ανθρώπων ε, για ανεξάρτητη διαβίωση. Αυτό σημαίνει να έχουμε τον έλεγχο της ζωής μας και να έχουμε την υποστήριξη που χρειαζόμαστε για να είμαστε ενεργά μέλη των κοινοτήτων μας. Ε, άλλωστε είμαστε και εμείς στοιχείο της ε, ανθρώπινης ποικιλομορφίας, αποκλειόμαστε όμως από την ε, κοινωνία. Εάν περπατήσετε ε, στους δρόμους των ευρωπαϊκών πρωτεύουσών ε, βλέπετε άτομα με αναπηρίες. Ε, όχι αρκετά, όχι αν λάβουμε υπόψη ότι είμαστε το 15% του πληθυσμού της Ευρώπης. Θα σας παρουσιάσω τις διαφάνειές μου, δεν θα τα διαβάσω όλα διότι περιέχουν πολλά στοιχεία. Θα ήθελα να αναφερθώ λοιπόν σε ένα συγκεκριμένο θέμα που μας έχει απασχολήσει, το άρθρο 19 Τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Ε, ο δικός μας σχολιασμός του άρθρου αυτού διευκρινίζει το άρθρο αυτό, διότι από τα 10 χρόνια εφαρμογής της Σύμβασης διαπιστώνουμε ότι ενώ φαίνεται το άρθρο να είναι σαφές, Η ερμηνεία του δεν είναι τόσο μονοσήμαντη όσο θα θέλαμε εμείς οι ακτιβιστέ για τα άτομα με αναπηρίε. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν ε, πρόσφατα ε, ασχολήθηκε με αυτόν τον γενικό σχολιασμό του άρθρου 19 που ασχολείται με την ανεξάρτητη διαβίωση και είναι πολύ σημαντικό αν σκεφτούμε θέματα νομικής και κοινωνικής προστασίας διότι είναι ένα θέμα το οποίο διέπει όλες τις πτυχές ε, της ε, ζωής των ε, ατόμων με αναπηρίες. Θα αναφερθώ λοιπόν σε τρία εμπόδια από τον μακρύ κατάλογο που έχουμε. Αυτό σχετίζεται με αυτό που είπε ο Βίλεμ. Έχει να κάνει με την νομική μας ικανότητα. Είναι σημαντικό τα άτομα με αναπηρίες να έχουν ε, λόγο όσον αφορά τη ζωή τους ε, και να μπορούν να ε, επιλέγουν. Πώς μπορεί να γίνει αυτό εάν κάποιος μας αρνηθεί την νομική ικανότητα. Οι μη ανάπηροι δεν χρειάζεται να δικαιολογήσουν κάθε κακή απόφαση που λαμβάνουν, αλλά για άτομα με αναπηρίες ε, μόλις ε, λάβουν μια κακή απόφαση αμέσως αμφισβητείται ε, η ικανότητά τους να λαμβάνουν αποφάσεις. Αυτή τη στιγμή πολύ μεγάλο μέρος της παρακολούθησης των συστημάτων προστασίας εξαρτάται από τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών όσον αφορά τη διαπίστωση εφαρμογής ε, των νόμων. Δυστυχώς υπάρχει μια αυξανόμενη τάση προς ιδρυματοποίηση. Τα ιδρύματα όμως δεν αποτελούν λύση και όμως σε εποχές λιτώσεις, λιτότητας ε, βλέπουμε να προωθούνται ακόμη τα ιδρύματα ως επιλογή. Και τα ιδρύματα δεν θα αποτελέσουν ποτέ σωστή επιλογή αν θέλουμε να λάβουμε υπόψη μας τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ένα από τα βασικά στοιχεία ε, της, ε, αυτού του γενικού σχολείου είναι να ζητήσουμε παρακολούθηση και επιβολή κυρώσεων όταν ε, δεν παρέχεται η βασική πρόσβαση σε βασικές ε, υπηρεσίες. Εάν ε, δεν υπάρχει πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, τότε αναγκάζεται κανείς στον αποκλεισμό. Οι περισσότεροι ε, τα περισσότερα άτομα με αναπηρίες χρειάζονται πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες ε, στις οποίες έχουν πρόσβαση τα άτομα χωρίς αναπηρίες. Ε, δεν χρειάζεται λοιπόν να υπάρχει δαπανηρή ξεχωριστή παροχή των υπηρεσιών αυτών. Επίσης θέλουμε περισσότερη χρηματοδότηση για την ανεξάρτητη διαβίωση όπου ε, οι υπηρεσίες παρέχονται χωρίς αποκλεισμούς. Τα άτομα με αναπηρίε αποτελούν μέρος της κοινωνίας και έχουμε πολλά να προσφέρουμε. Εάν λοιπόν απομονωθούμε ε, και δεν έχουμε ανεξάρτητη διαβίωση δεν μπορούμε να συμβάλλουμε στις κοινωνίες μας ε, στο μέτρο του δυνατού. θα πρέπει να υπάρχει υποχρέωση εξάλληψης των εμποδίων ε, στην ε, πρόσβαση υπηρεσιών, διότι αν δεν εξαλείψουμε αυτά τα εμπόδια, αυτό θα είναι όλο και πιο δαπανηρό στο μέλλον. Θα πρέπει να φροντίσουμε τα άτομα με αναπηρίες και οι οργανώσεις μας να συμμετέχουν ενεργά στην λήψη αποφάσεων ε, που σχετίζονται με τις υπηρεσίες για να μπορούμε να έχουμε υπηρεσίες χωρίς αποκλεισμούς και προσβάσιμες από όλους. Δεν θα πρέπει να δαπανώνται δημόσιοι πόροι για την ε, διατήρηση ιδρυμάτων ε, κανενός τύπου ή οδήποτε τύπου. Βλέπουμε ότι σε διάφορες χώρες ε, τα διευθυντικά ταμεία χρησιμοποιούνται για την πρόθεση και ανάπτυξη ιδρυμάτων. Αυτό όμως ε, δεν γίνεται στο πνεύμα της ε, σύμβασης ε, του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, ούτε βελτιώνει το επίπεδο διαβίωσης των ατόμων με αναπηρίες. Μία από τις προϋποθέσεις που χρειαζόμαστε για να μπορούμε να ολοκληρώσουμε την κοινωνική προστασία είναι η πρόσβαση σε πληροφορίες, διότι υπάρχουν πολλοί τύποι προστασίας. Αυτή τη στιγμή όμως πρέπει να έχει κανείς στοιχείο νομικής για να μπορεί να επωφεληθεί από αυτούς τους τύπους προστασίας. Χρειαζόμαστε λοιπόν προσβάσιμες πληροφορίες ώστε να μπορούμε να επωφεληθούμε από τα διάφορα είδη προστασίας. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει πρόσβαση στη δικαιοσύνη χαμηλού κόστους ώστε ε, να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους μηχανισμούς που υπάρχουν και θα πρέπει να φροντίσουμε ε, να υπάρχει διαβούλευση με τους ανθρώπους αυτούς ε, κατά την εκπόνηση των μηχανισμών. Δεν έχει νόημα να υπάρχουν μηχανισμοί που απαιτούν από άτομα με αναπηρίε ή από άλλου φορεί να ταπανούν ένα σωρό χρήματα, ενώ αυτό δεν είναι απαραίτητο. Θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ε, ότι η επιλογή και ο έλεγχος αποτελεί τη βάση για όλα όσα κάνουμε. Είναι ο λόγος που αγωνιζόμαστε για την ανεξάρτητη διαβίωση εάν μπορεί κανείς να έχει έλεγχο και επιλογή στη ζωή του εάν δεν γνωρίζει τι ε, προστασία του παρέχεται και πώς λειτουργεί το σύστημα. Αυτή τη στιγμή τα άτομα με αναπηρίε αναμένεται να γνωρίζουν πολύ περισσότερα από τον μέσο πολίτη σχετικά με νομικούς μηχανισμούς για να έχει πρόσβαση ε, σε υπηρεσίες ε, οποία, σε οποίες έχει αυτόματη πρόσβαση ένας άνθρωπος χωρίς αναπηρίες. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας ε, και αν υπάρχουν ερωτήσεις πολύ ευχαριστώ θα απαντήσω. Ευχαριστώ πολύ κυρία Τόντ και εσείς ε, τηρήσατε απόλυτα το δεκάλεπτο και τώρα να δώσω το λόγο στον τελευταίο ομιλητή, στον κύριο Τόμας Πινιάλ. Παρακαλώ έχετε το λόγο. Uh, Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να μιλήσουμε σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ ε, σημαντική συνεδρίαση σε αυτό το εργαστήριο. Ο τίτλος ήταν «Νομική και κοινωνική προστασία των ατόμων με αναπηρία» και οι πρώτες μου σκέψεις όταν, άκουσα το, όταν διάβασα τον τίτλο είναι ότι θα πρέπει να δούμε τη νομική και κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία. Ο όρο προστασία ίσω επινοήθηκε κάποια στιγμή που προσπαθούσαμε να φροντίσουμε τα άτομα με αναπηρία αντί να προσπαθούμε να τα εντάξουμε στην κοινωνία και παρά το γεγονό ότι ε, η ένταξη σημαίνει και προστασία και πρέπει να προστατεύονται, είναι πολύ σημαντικό να εντάσσονται και στην κοινωνία και αυτό ίσω θα μπορούσε να αποτελέσει και τροχή για, προφή σκέψη για τη συνέχεια τη παρουσίασή μου. Ποιοι είμαστε. Εργάζομαι για μια διαφορετική οργάνωση σε σχέση με αυτή που μίλησαν προηγουμένω. Αναφέρομαι στι ε, ε, υπηρεσίε φροντίδα και στήριξη των ατόμων με αναπηρία. Είμαστε γνωστοί με τα αρχικά EASPD. Εκπροσωπούμε περίπου 15.000 υπηρεσίε φροντίδα και στήριξη σε 33 διαφορετικέ χώρε και εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και παρέχουμε φροντίδα, παιδεία, απασχόληση κλπ. Είμαστε βασικό βασικός τη Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεργαζόμαστε με του φίλου μα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με του φίλου μα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά επίση συμμετέχουμε και στο Συμβούλιο τη Ευρώπη και στα Ηνωμένα Έθνη, που είμαστε ε, διαπιστευμένα μέλη ε, των κοινωνικών μερών και φυσικά ε, συνεργαζόμαστε και με του συναδέλφου εδώ στι Βρυξέλλες που εκπροσωπούν και αυτοί άτομα με αναπηρίε και άλλε μη κυβερνητικέ οργανώσει. Ποιο είναι ο στόχο μα, θέλουμε να προωθήσουμε αποτελεσματικές ε, και ε, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και συστήματα. Ακούσαμε σήμερα ότι υπάρχουν ακόμα θεσμικά όργανα που κάνουν ε, διακρίσεις ε, στα άτομα με αναπηρία. Ειδικά σχολεία που και πάλι κάνουν διάκριση ε, στα άτομα με αναπηρία και αποκλείουν άτομα από τα εκπαιδευτικά συστήματα. Εμείς εκπροσωπούμε ένα τομέα ο οποίος παρέχει αυτές τις υπηρεσίες αλλά ταυτόχρονα συμμετέχει ενεργά για να υπάρξει μια εξέλιξη και αλλαγή και να συνάδουν περισσότερο με τα όσα προτείνεται από την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών. Όλα μας τα μέλη συμμετέχουν ενεργά σε συζητήσει συζητήσεις, διαπραγματεύσει, ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών για το πώ μπορούμε να υποστηρίξουμε με τον καλύτερο τρόπο τα άτομα με αναπηρία δεδομένων των δομών που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή. Και προσπαθούμε φυσικά να δεσμευτούμε στον τομέα αυτό. Τα άτομα με αναπηρία πρέπει να έχουν ε, συστήματα υποστήριξη υψηλή ποιότητα, να υπάρχει ίση πρόσβαση σε υγεία, σε εκπαίδευση, απασχόληση, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον και να ζουν ανεξάρτητα και να έχουν την ελευθερία να κάνουν τι ε, προσωπικέ του επιλογέ. Και πώς γίνεται αυτό. Εργαζόμαστε σε διάφορους τομείς. Εγώ θα επικεντρωθώ σε ελάχιστους εξ αυτών. Ε, εργασία απασχόληση. Παρέχονται υπηρεσίες απασχόλησης, ε, επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας ε, και υπάρχουν και εργαστήρια διαφόρων μορφών. Προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία ε, των μελών μας και τις γνώσεις τους για να δώσουμε συμβουλές και συστάσεις στους ηθήνοντες πολιτικής... για το πώς πρέπει να χαράσουν οι πολιτικές. Για παράδειγμα, εργαστήκαμε στην εγγύηση για την νεολαία. Πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ σημαντική ευρωπαϊκή ε, πολιτική έχει πρόσβαση για τα άτομα αναπηρία. Σε κάποιες χώρες όχι. Στην Ιρλανδία, για παράδειγμα, για να συμμετέχει κάποιο στην εγγύηση για την νεολαία θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένο στο βασικό μητρό, αλλά είναι αν είσαι άτομο με αναπηρίο και παίρνει επίδομα αναπηρία, δεν μπορεί να εγγραφεί στο Μητρό, επομένω δεν μπορεί να συμμετέχει ενεργά στην εγγύηση για την νεολαία. Και αυτό είναι σαφώ πρόβλημα. Υπάρχουν επίση κάποιε περιπτώσει ε, μακροπρόθεσμη στήριξη και βοήθεια ε, στα άτομα με αναπηρία για να παραμείνουν στη θέση εργασία του αφού αποκτήσουν και την κατάλληλη επαγγελματική εμπειρία μέσω τη εγγύηση για την νεολαία. Και θέλουμε να το προωθήσουμε και αυτό. Επίσης, ασχολούμαστε και με εκθέσεις πολιτικής. Προσφάτως δημοσιεύτηκε και μία έκθεση η οποία καταδεικνύει ότι η δημόσια χρηματοδότηση και η βοήθεια προς τους ανθρώπους για τα, ε, σε να αποκτήσουν θέσεις εργασίας ε, είναι πιο φθηνή μορφή για τους φορολογουμένους. Επομένως, ε, θέλουμε να στηρίξουμε τα άτομα με αναπηρία για να βρεθούν στην αγορά εργασίας, ε, βέβαια για τους λόγους ε, που αναφέρονται και για τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, τα δικαιώματα, τις αξίες κλπ. Αλλά και γενικότερα για τον πληθυσμό, δεδομένου ότι έχουμε και μια γυράσκουσα κοινωνία. Υπάρχουν άτομα τα οποία ε, είναι ειδικά σχολεία, σχολεία ειδική αγωγή, ε, σχολεία που προσπαθούν να περιλάβουν του πάντε και προσπαθούμε να πάνε όλα τα σχολεία προ ε, μία εκπαίδευση χωρί αποκλεισμού και φυσικά χρηματοδοτούνται και πάρα πολλά προγράμματα τα οποία έχουν στόχο να μα υποστηρίξουν σε αυτή τη διαδικασία. Ε, το να ζει κάποιο ανεξάρτητα και να υπάρχουν συγκεκριμένε κοινωνικέ υπηρεσίε. Υπάρχουν ε, δομέ στην Ευρώπη, αλλά υπάρχουν αρκετέ εκκρεμότητε. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα ξεφύγουμε από αυτή την παρεχημένη διαδικασία για να έχουμε υπηρεσίε που βασίζονται στην κοινότητα και φυσικά αυτό χρειάζεται και κατάλληλε πολιτικέ. Γι' αυτό συνεργαζόμαστε και με τα ευρωπαϊκά όργανα, αλλά και με του συναδέλφου από αντίστοιχε οργανώσει. Και φυσικά έχουμε και άλλα σημαντικά θέματα. Ακούσαμε προηγουμένω την εκπαίδευση χωρί αποκλεισμού και πόσο μπορούμε να τα συμπεριλάβουμε όλα αυτά. Και φυσικά όλα αυτά έχουν σημασία και από πλευρά αξιών και πρέπει να αναγνωρίσουμε όμω και ότι όσο νωρίτερα αποκλειστεί ένα άτομο με αναπηρία από την κοινωνία, τόσο πιο δαπανηρό γίνεται για την κοινωνία. Γιατί πρέπει να υποστηρίξουμε έναν άνθρωπο ο οποίο έχει ζήσει αποκλεισμένο όλη του τη ζωή για να τον βοηθήσουμε να βρει μια θέση εργασία ε, στο μέλλον. Θα πρέπει να το εξετάσουμε και αυτό και από αυτό το πρίσμα. Επίση, νέε τάσει, νέε τεχνολογίε, πώ μα βοηθούν να παρέχουμε καλύτερε υπηρεσίε. Ε, όχι μόνο για τα άτομα με αναπηρία, αλλά γενικότερα ο τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών για καλύτερη στήριξη των ηλικιωμένων ατόμων. Ασχολούμαστε και με αυτά. Ε, τέχνες, αθλητισμός, ε, στήριξη για συμμετοχή σε αυτά, συμμετοχή στον πολιτισμό, σε αθλητικές δραστηριότητες και φυσικά μας βοηθούν και τα ευρωπαϊκά κονδύλια εδώ. Ένα άλλο θέμα το οποίο μας απασχολεί πολύ ε, είναι ο τομέας των κοινωνικών υπηρεσιών που είναι ο μεγαλύτερος αυτή τη στιγμή, δημιουργεί τις περισσότερες θέσεις εργασίας, πάνω από 1,7 εκατομμύριο θέσεις εργασίας τα τελευταία χρόνια ε, φροντίδα παιδιών, φροντίδα ατόμων με αναπηρία, υποστήριξη ατόμων με αναπηρία. Αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό και επίση υποστήριξη ηλικιωμένων ατόμων για να μπορούν να ζουν ε, μια ζωή ανεξάρτητη. Ε, δημιουργούμε αυτέ τι θέσει εργασία, αλλά το πρόβλημα είναι ότι κανεί δεν θέλει να κάνει πια αυτές τις Υπάρχουν πιέσει και για τη δημόσια χρηματοδότηση, αλλά όχι μόνο αυτό. Ε, υπάρχει λοιπόν ε, κακοπληρωμή σε αυτές τις δουλειές ε, και ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται. Πολλοί νέοι άνθρωποι προτιμούν να εργαζόνται σε ένα σούπερ μάρκετ αντί στι υπηρεσίε φροντίδε. και αυτό είναι πρόβλημα και γι' αυτό ακριβώ και προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι ο τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών θα είναι τμήμα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Διαλόγου. Δεν μπορεί να μην εκπροσωπούνται αυτέ οι υπηρεσίε και να σα πω ότι την επόμενη εβδομάδα θα εξηγήσει ε, μια νέα ομοσπονδία εργοδοτών που θα λέγεται Ομοσπονδία Κοινωνικών Εργοδοτών που θα προσπαθήσουν να βρουν λύσει για ελλείψει σε προσωπικό, πρόσληψη και προσοχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να αντιμετωπίσουμε και τα θέματα αυτά και φυσικά ε, να μπορέσουμε να πιέσουμε και τα θεσμικά όργανα. Επίσης, ε, το θέμα των μεταναστών με αναπηρίες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα ε, συμφώνησε να χρηματοδοτήσει ένα πρόγραμμά μας για να ε, φέρουμε σε επαφή μετανάστες με αναπηρία ε, με τις υπηρεσίες που χρειάζονται και τις δομές στήριξης στην Ελλάδα και στις άλλες ενοριακές χώρες αλλά και στη Φιλανδία, τη Γερμανία και στην Αυστρία σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης κλπ. Προσπαθούμε ε, και με τις πιο εξειδικευμένες δομές και υπηρεσίες ε, προσπαθούμε να γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Και έχουμε και οριζόντια θέματα συμπαραγωγή, πώς μπορούμε να έχουμε συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία για να αποφασίσουν πώς θέλουν να οργανώνονται οι υπηρεσίες και η στήριξη που τους παρέχεται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και νέοι τρόποι χρηματοδότησης των υπηρεσιών. Είναι πολύ καλά τα διορθωτικά τομέα στον τομέα αυτό. Υποστηρίζουν τη μετάβαση σε υπηρεσίες βάσει της κοινότητας. Ε, πολλά πράγματα για το σχέδιο Juncker, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, για να έχουμε καλύτερη πρόσβαση ε, και κατασκευή νέων κοινωνικών υποδομών, για να μπορέσουμε να άρουμε κάποιους από τους φραγμούς εκεί και φυσικά κρατικές προμήθειες ε, και ενισχύσεις. Τι μέλη γενέστε. Δεν είναι εύκολο το θέμα αυτό να το συζητήσουμε. Ε, πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία των βασικών ε, ενδιαφερομένων. Πρέπει να βρεθεί το θέμα αυτό στο επίκεντρο της διαδικασίας χάραξης πολιτικής. Τις προάλλες είδα μια παράθεση που έλεγε ότι δεν υπάρχει ε, Τρόπο να αποφύγουμε την ειρήνη, η ειρήνη είναι η λύση και εγώ θα το παραφράσω και θα πω δεν υπάρχει τρόπος να αποφύγουμε την ένταξη, η ένταξη είναι η λύση. Είναι πάρα πολύ καλός τρόπος λοιπόν να προχωρήσουμε, πρέπει να δούμε πώς θα τα εφαρμόσουμε αυτά στην πράξη και θα τα συμπεριλάβουμε παντού. Επίσης πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να ε, εξορθρολογήσουμε, δεν μπορούμε να έχουμε μια ε, κοινωνία που περιλαμβάνει τους πάντες εάν ε, δεν υπάρχει συνεργασία με τα άτομα με αναπηρία. Πρέπει να συνεργαστούμε με του τους εργοδότες, με τις τοπικές αρχές. Ε, όλοι εδώ ε, είναι ειδικοί σε θέματα αναπηρίας, επικεντρώνονται σε αυτό και είναι πολύ σημαντικό, αλλά είναι πολύ σημαντικό να συνεργαστούμε και με άλλους ενδιαφερομένους. Ε, πρέπει να αναπτύξουμε γνώσεις και πυρογνωμοσύνη, έλλειψη δεδομένων πολύ συχνά, κυρίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και για τα άτομα με αναπηρία, αλλά και για τις κοινωνικές υπηρεσίες. Δεν υπάρχουν στοιχεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο που να γνωρίζουν πόσα δημόσια κονδύλια πηγαίνουν στις κοινωνικές υπηρεσίες στην Ευρώπη. Δεν ξέρουμε πώ έχουν εξελιχθεί αυτά στην τελευταία δεκαετία και πρέπει να το εξετάσουμε. Και τέλος, από πλευράς μας ως ε, πάροχοι κοινωνικών υπηρεσιών πρέπει να ε, αλλάξουμε νοοτροπία και να μην σκεφτόμαστε ότι η βοήθεια στα άτομα με αναπηρία είναι κόστος. Είναι επένδυση. Πρέπει να το σκεφτόμαστε τελείως διαφορετικό, κυρίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Μπίγναλ. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές για τη συμμετοχή τους, όπως είπα και πριν. Έχετε την δυνατότητα να θέσετε ερωτήσεις ή ε, κάποια σχόλια, είτε από πλευράς βουλευτών, είτε από πλευράς ε, προσκεκλημένων. Δεν ξέρω αν κάποιος θα ήθελε το λόγο. Ε, ήταν σαφής οι παρεμβάσεις σας από ό,τι φαίνεται και πληρέστατες και εφόσον λοιπόν δεν υπάρχουν περαιτέρω ερωτήσεις θα ήθελα να κλείσω λοιπόν το τμήμα αυτό του workshop να ευχαριστήσω όλους όσους πήραν μέρος στις εργασίες και κατέστησαν ε, το τμήμα αυτό της συνεδρίασης ε, ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Θα δώσω το λόγο τώρα στην πρόεδρο κυρία Βίκστρομ για τα υπόλοιπα θέματα ε, με συγκεκριμένες αναφορές τις οποίες αναφέρθηκα στην αρχή ε, δηλαδή τα θέματα τα οποία συζητήσαμε μέσω συγκεκριμένων περιπτώσεων αναφορών. Σας ευχαριστώ και εγώ εξ ονόματος της Επιτροπής θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους εσάς που πήρατε μέρος σήμερα το πρωί σε μια καρποφόρα ανταλλαγή απόψεων. Φυσικά αυτά που ακούσαμε είναι πάρα πολύ χρήσιμα όπως και τα έγγραφα τα οποία μας προτείνεται. Είναι κάτι το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε ε, όχι μόνο εμείς στην Επιτροπή Αναφορών αλλά και άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές στο Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους για την συνεισφορά σας. Σας εύχομαι καλή συνέχεια. Θα συνεχίσουμε τον διάλογο τις επόμενες μέρες. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στα υπόλοιπα θέματα. Θα ήθελα να καλωσορίσω τώρα τον Edward Deering, ο οποίος ε, είναι μαζί μας μαζί με τη Laura Lear, και τον Αλεξάνδρ Μακρύμπ. Σας καλωσορίζω, έχετε το λόγο για την 1305 ε, προβλήματα ανθρώπων με αναπηρίες που δεν ενημερώνονται σωστά από τις αρμόδιες αρχές στην ε, Ιρλανδία. Έχετε το λόγο κύριε Ντίρινγκ. Κοιτάξτε, ο κύριος Ντίρινγκ είναι εδώ για να σας παρουσιάσει την αναφορά του και θα διαβάσω την αναφορά αυτή εγώ εκ μέρους του. Έχει σοβαρή δυσλεξία και οι υπηρεσίες γεωργίες δεν τον βοήθησαν να κατανοήσει και να εφαρμόσει τους κανόνες σε σχέση με την γεωργία γενικότερα τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την οδηγία για την έλογη χρήση ζυζανιοκτώνων. Χρειάζεται λοιπόν σωστή ενημέρωση για να ασκήσει τις ευθύνες του, τις υποχρεώσεις του, αλλά δυστυχώς οι αρμόδιες Ιρλανδικές υπηρεσίες απέτυχαν. Όταν ήρθε σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Ένωση ενημερώθηκε ότι τα κράτη-μέλη έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν σωστά τους πολίτες που ε, είναι δικαιούχοι ε, κοινοτικών πιστώσεων. Αυτό δεν έγινε στην περίπτωση του. Ε, ταυτόχρονα ε, θα έπρεπε οι πληροφορίες να του δοθούν σε κατανοητή μορφή. Αυτό για πολλά χρόνια ε, διαμαρτύρεται ο κύριος Ντίρινγκ ότι δεν έχει αλλάξει. Ο κύριος Ντίρινγκ θέλει να μπορέσει να είναι πραγματικά ικανός να καλλιεργήσει τα εδάφη του, αλλά δυστυχώς δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα και οι διαχειριστικές αρχές στην Ιρλανδία δεν φέρουν εις πέρα στις υποχρεώσεις τις οποίες έχουν. Νομίζω ότι η Εθνική Αρχή Αναπηρίας της Ιρλανδίας ενημέρωσε και σας ενημέρωσε και εσάς ότι υπάρχουν οι λεγόμενοι access officers, υπεύθυνοι πρόσβασης ε, ρόλος τους είναι να βοηθούν ακριβώς τους πολίτες που έχουν ε, προβλήματα να κατανοούν σημαντικές πληροφορίες, νομοθετικές πληροφορίες κτλ. Σαν παράδειγμα ένας άνθρωπος με τις δυσκολίες ε, του κυρίου Ντίρινγκ πρέπει να του διαβάζουν τους κανόνες ή να τους τις δίνουν μαγνητοφωνημένες. Δυστυχώς όμως οι υπηρεσίες και οι υπεύθυνοι για την πρόσβαση δεν το έχουν κάνει αυτό και δεν μπορεί ακριβώς σαν παράδειγμα να είναι συμβατές οι πρακτικές του με την οδηγία για την σωστή χρήση των ζυζανιοκτώνων. Θα έπρεπε στα πλαίσια της οδηγίας αυτής να πάρει κάποια πιστοποίηση, αλλά δεν είναι σε θέση να το κάνει αυτό και δεν του δόθηκαν εναλλακτικές λύσεις. Η αποτυχία αυτή ε, να μπορέσει δηλαδή ε, δυστυχώς του στερούν την δυνατότητα να συνεχίσει να καλλιεργεί τη γη του. Είχε προβλήματα εξ αρχής ε, στην γραφή και στην ανάγνωση και μόνο όταν ενηλικιώθηκε έμαθε ότι υποφέρει από μια πολύ σοβαρή δυσλεξία και αυτό είναι κάτι το οποίο δυστυχώς του στερεί τη δυνατότητα να καλλιεργήσει το έδαφος το οποίο έχει στην κατοχή του. Είναι συστηματική πλέον η αποτυχία του Υπουργείου Γεωργίας της Ιβλανδίας να τον βοηθήσει αυτόν και τους συναδέλφους του με αντίστοιχες δυσκολίες. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας ευχαριστήσει ο κύριος Ντίρινγκ και να σας ζητήσει παρακαλώ να συνεχίσετε να, να κρατάτε ανοιχτή την συγκεκριμένη αναφορά έτσι ώστε να υπάρξει προσβάσιμη και κατανοητή ενημέρωση από πλευράς των διαχειριστικών αρχών της χώρας του. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ντίριν και σας ευχαριστώ για την ανάγνωση που μας βοηθήσατε δηλαδή. Να γνωρίζουμε πλέον τις απόψεις σας γύρω από το θέμα αυτό. Θα στραφώ τώρα προς τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και να του δώσω το λόγο για να μας εξηγήσει τις θέσεις της υπηρεσίας του. Σας ευχαριστώ πολύ. Πράγματι πήραμε την ανακοίνωση του κυρίου Ντίρινγκ. Ανησυχούμε από το ότι η κατάσταση αυτή της δυσκολίας προσβασιμότητας, όπως λέει στην δήλωσή του, τον εμποδίζει από το να φέρει σφαίρα στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Η σοβαρή δυσλεξία είναι κάτι το οποίο πράγματι μπορεί να παρεμποδίσει την πρόσβαση στην πληροφόρηση. Είμαστε όμως βέβαιοι ότι μπορεί να βρεθούν λύσεις για να υποστηριχθούν οι άνθρωποι αυτοί να ενημερωθούν σωστότερα έχουν ε, ξεκινήσει και σε εθνικό επίπεδο κάποιες δράσεις οι οποίες δεν έχουν λύσει όμως το πρόβλημα του κ. Ντίρινγκ. Θα πρέπει να υπογραμμίσουμε πάντως ότι σχετικά και με τα διαφθρωτικά ταμεία Οι ενέργειες οι οποίες ε, μας απασχολούν εδώ αναφέρονται στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο και η επιστολή απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπογραμμίζει τον ρόλο της διαχειριστικής αρχής έτσι ώστε οι πολίτες δικαιούχοι των ταμείων να έχουν στη διάθεσή τους τις κατάλληλες πληροφορίες για την εφαρμόσιμη νομοθεσία. Όμως αυτό το οποίο θα ήθελα επιπλέον να πω είναι ότι λόγω της ανησυχίας αυτής λαμβάνουμε το θέμα αυτό πολύ σοβαρά και έχουμε κάνει κάποια βήματα για τη βελτίωση της κατάστασης. Να πω ότι στον κανονισμό της επόμενης προγραμματικής περίοδου 14-20 υπάρχουν πολύ περισσότερες προβλέψεις οι οποίες είναι σχετικές με τα θέματα της πρόσβασης ε, των ε, δικαιούχων στην ενημέρωση και ε, το παράρτημα 12 εδώ για τη σωστή ενημέρωση των δικαιούχων των διαφθορτικών ταμείων και τη σωστή περιγραφή του υλικού που είναι απαραίτητη. Λοιπόν, εμείς θα καταστήσουμε προσβάσιμα τα έγγραφα αυτά και τις πληροφορίες αυτές για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί μέχρι τώρα λυπούμεθα, αλλά νομίζω ότι θα συνεχίσουμε την προσπάθεια να βελτιώσουμε την προσβασιμότητα όχι μόνο στο θέμα της ε, βελτίωσης πρόσβασης στην ενημέρωση αλλά γενικότερα. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Η Ρώσα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς ε, να ευχαριστήσω τους αναφέροντες. Είναι ένα παράδειγμα ε, διότι πριν ακριβώς ε, από τις αναφορές αυτές είχαμε ένα εργαστήριο και έχουμε αυτή την αναφορά του συναδέλφου από την Ιρλανδία όσον αφορά τη δυσκολία πρόσβασης σε ε, πληροφορίες σε μορφή προσβάσιμη για τα άτομα με αναπηρία. Πρόκειται για ένα παράδειγμα, μια πολύ σοβαρή μορφή δυσλεξίας, ε, η διάγνωση ήρθε ε, αρκετά καθυστερημένα και αυτή τη φορά το Υπουργείο Γεωργίας δεν παρέχει προσβάσιμες πληροφορίες και αυτό αποτελεί διάκριση για την ζωή του αναφορεμένου. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά. Η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν απόλυτα σαφής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί ε, να υπάρχει πραγματική προσβασιμότητα. Γι' αυτό ακριβώ και θα ήθελα να προτείνω να μπορούμε να αποτανθούμε και στην κυβέρνηση της Ιρλανδίας, στο Υπουργείο Γεωργίας, και να ζητήσουμε πληροφορίες για να μην επαναληφθεί ε, ε, ένα τέτοιο θέμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι πληροφορίες να είναι σε μορφή προσβάσιμη. Αλλιώς υπάρχει σαφής ε, διάκριση για τις ίσες ευκαιρίες των ατόμων και σε αυτή την περίπτωση για τα άτομα με αναπηρία. Και νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να αποτανθούμε στις αρχές, και επίση και στην Εθνική Αρχή αναπηρία και στο Υπουργείο Γεωργία τη Ιρλανδίας για να ε, μπορέσουν να μας ε, ε, πούνε για την πρόσβαση των πληροφοριών, να φροντίσουν να είναι προσβάσιμες οι πληροφορίε και οι παρούσε και οι Ευχαριστώ κυρία Νεριάντα, καλωσορίσατε στην επιστροφή, δεν σα έχω ξαναδεί, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να λάβω το λόγο. Θα είμαι σύντομη. Είμαι εδώ για να υποστηρίξω τον κύριο Ντίρινγκ και να ευχαριστήσω και τον Μπράιν Κρόλι που εκπροσωπείται εδώ και υποστηρίζει και τον κύριο Ντίρινγκ ένα-δυο σχόλια. Πραγματικά πιστεύω ότι τη σήμερα ημέρα δεν είναι δυνατόν. Υπάρχει τεχνολογία, μπορεί να υπάρχουν οπτικοακουστικές υπηρεσίες διαθέσιμες. Είναι πολύ απλό, δεν χρειάζεται να επινοήσουμε τον τροχό γι' αυτό, ιδιαίτερα όταν αναφερόμαστε στη δυσλεξία. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Πρέπει να ασκήσουμε πιέσει στι τοπικέ αρχέ να παρέχουν αυτέ τι πληροφορίε στον κύριο Ντύριν και σε οποιονδήποτε άλλο έχει δυσλεξία. Και επίση πρέπει να πω ότι είναι ένα ευρύτερο θέμα. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα διάγνωση σε πολύ μικρότερη ηλικία. Αυτό είναι αποτυχία του εκπαιδευτικού συστήματο και ένα ακόμα σχόλιο το οποίο θα ήθελα να κάνω. Με τον τρόπο με τον οποίο προχωρούν τα πράγματα και φαντάζομαι ότι αντίστοιχα πράγματα συμβαίνουν και στα κράτη-μέλη, δεν υπάρχει πλήρη πρόσβαση σε βριζονικέ υπηρεσίε. Υπάρχουν μεγάλα τμήματα στην Ιρλανδία που δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο και πολλοί από τους κανόνες και τις κανονισμούς πρέπει να εφαρμόζονται διαδικτυακά και πρέπει να γίνονται απευθείας τα άτομα τα οποία δεν έχουν γνώσει υπολογιστών ή δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι εντελώ αποκλεισμένα. Στην περίπτωση του κυρίου Ντίρινγκ, το γεγονό ότι δεν μπορεί να καλλιεργήσει τη γη του είναι κατάφορη παραβίαση των δικαιωμάτων του. Πρέπει να μπορεί να καλλιεργήσει τη γη του, πρέπει να υπάρξουν πιέσει και πρέπει να το βρούμε και ένα χρονικό όριο γι' αυτό γιατί έχει καθυστερήσει η κατάσταση. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πιέσει τι ε, τοπικέ αρχέ, να παρέχουν αυτέ τι οπτικοακουστικές υπηρεσίε που είναι απαραίτητε για τον κύριο Ντίρινγκ. Καλή επιτυχία και ελπίζω να ξαναέρθω σύντομα στην Επιτροπή Αναφορών. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πάντα όταν κάποιο παίρνει το λόγο για πρώτη φορά στην Επιτροπή μα ε, και λέει τόσο σημαντικά πράγματα. Εξαιρετικό αυτό. Ε, οι νέε τεχνολογίε πληροφορική ε, είναι το κλειδί και ουσιαστικά από άγνοια δεν έχουν εφαρμοστεί μέχρι τώρα. Όπως είπατε, δεν ε, χρειάζεται να παρεφεύγουμε τον τροχό, χρειάζεται να εργαστούμε πάνω σε κάτι που ήδη υπάρχει και να είναι διαθέσιμο σε όλους. Είναι θέμα προσβασιμότητας. Ποιος άλλος θα ήθελε να πάρει το λόγο. Ο κύριος Μαριάς, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, για την ε, αναφορά 1305 είχαμε ζητήσει να ε, μπει ως ε, κατεπίγουσα στη συζήτηση. Αυτό δεν είναι. Και αυτή είναι μια αναφορά την οποία έθελε να υποστηρίξει ο συνάδελφός μου ο κύριος Κράουλη, ο οποίος βεβαίως ε, δεν έχει την δυνατότητα αυτή. Ε, με παρακάλεσε λοιπόν να ζητήσω να επισπευστεί η διαδικασία. Θεωρώ σημαντικό και να ευχαριστήσω την Επιτροπή που έκανε δεκτό το αίτημα να συζητηθεί σήμερα αυτή η αναφορά και θεωρώ ότι θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή. Είναι μια κλασική περίπτωση ε, σύμφωνα με την οποία οι πληροφορίες που λαμβάνει ένα άτομο με ειδικές ανάγκες από μια ανεξάρτητη αρχή δεν ήταν τέτοιες ε, που να μπορέσει ο ίδιος ως άτομο με ειδικέ ανάγκες να αντιληφθεί τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και το τι περιείχε αναλυτικά ο κανονισμός. Ως εκ τούτου του επευλήθη ένα πρόστιμο ε, που νομίζω ότι εάν δεν είχε αυτά τα προβλήματα ο ίδιος ε, θα μπορούσε υπό normal συνθήκες να έχει αντιληφθεί τι έπρεπε να κάνει και πώς να ακολουθήσει τους κανονισμούς που έχουν σχέση με την κοινή αγροτική πολιτική. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να μείνει ανοιχτή η υπόθεση αυτή. Θα πρέπει να ζητηθεί από την ανεξάρτητη αρχή στην Ιρλανδία να μην του επιβληθεί αυτό το πρόστιμο και να είναι και αφορμή αν θέλετε και σε επίπεδο Ιρλανδίας αλλά και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη οι αρμόδιες αρχές που χειρίζονται τέτοια θέματα όταν έχουν ζητήματα επικοινωνίας και ενημέρωσης σε άτομα με ειδικέ ανάγκες να έχουν μια διαφορετική προσέγγιση. Νομίζω ότι οι εισηγήσει που έγιναν το πρωί παρακολούθησα λίγη ώρα ορισμένες από αυτές γιατί όφυλα να είμαι και σε άλλη επιτροπή δυστυχώς ε, ε, ανέδειξαν όλο το ζήτημα και ευτυχώς που υπάρχει το live streaming και ε, γίνεται γνωστό όλο ε, γνωστό, ε, όλο γνωστός όλος αυτός ο προβληματισμός. Επομένως, ε, συμφωνώ και εγώ με την πρόταση να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά, να επικοινωνήσουμε με τις αρχές στην Ιρλανδία και να κυρίως να σταματήσει το πρόστιμο το οποίο υπάρχει εις βάρος αυτού του προσώπου του petitioner από την Ιρλανδία, ο οποίος μάλιστα δεν απευθύνθηκε καν μόνος του, αλλά ζήτησε και τη συμπαράσταση ενός συναδέλφου ε, ε, που είναι στην Ιρλανδία και ο οποίος και αυτός αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα υγείας. Σας ευχαριστώ πολύ. I thank you. Ευχαριστώ εγώ. Κύριε Ντίερινγκ, θέλετε να κάνετε κάποιες τελευταίες παρατηρήσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που άκουσε την υπόθεσή μου και θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, τον Brian Crowley και ε, και τον Liam Μουέρτε που ανέλαβε την υπόθεσή μου και ε, ελπίζω να καταλήξουμε σε καλό αποτέλεσμα. Πρόεδρος. Ε, ντροπή θα ήταν ε, εάν ε, δεν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα αφού κάνατε τον κόπο να έρθετε στις Βρυξέλλες να υποβάλλετε αναφορά και να ασχοληθείτε με το θέμα αυτό για τόσο καιρό. Ήρθατε εδώ πέρα μαζί με τους φίλους σας. Νομίζω ότι είσαστε ήρωας. So, thank you σας, ευχαριστώ θερμά που ήρθατε και που μας μεταφέρατε το μήνυμά σας. Πιστέψτε με, έχουμε εξετάσει πολύ σοβαρά την αναφορά σας και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ καλό παράδειγμα όπου θα είναι η απαραίτητη η αυξημένη διοργανική συνεργασία για να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Και να σας αναφέρω τι θα κάνουμε εδώ στην Επιτροπή μας. Φυσικά θα παραμείνει ανοιχτή η αναφορά. Θα στείλουμε επιστολή στο ε, Ιρλανδικό Υπουργείο Γεωργίας όπου θα ζητάμε την ε, γνώμη τους για την προσβασιμότητα σε πληροφορίες που παρέχει το Υπουργείο σε, από άτομα ε, με σοβαρή δυσλεξία καθώς και την βοήθεια που μπορεί να παρέχεται στις περιπτώσεις αυτές και τονίσουμε την ύπαρξη νέων τεχνολογιών, θα τονίσουμε την ύπαρξη της ε, πράξης για την προσβασιμότητα και θα τους πούμε ότι ειλικρινά ζούμε στον 20ο αιώνα, 21ο αιώνα, συγγνώμη, και οι αρχές θα πρέπει να προσαρμοστούν στα δεδομένα του νέου αιώνα. Να παρέχουν τις πληροφορίες με τρόπο φιλικό προς ε, τον χρήστη. Αυτά μπορούμε να κάνουμε Κύριε Μαριά, έχετε να προσθέσετε κάτι. Καταρχά, όπω και εσείς ε, είπατε, να συγχαρούμε τον ε, αναφέροντα για την τεράστια προσπάθεια που έκανε και να είναι εδώ. Όμως, επειδή του έχει επιβληθεί και πρόστιμο, θα πρέπει κατά την άποψή μου να υπάρχει μια αναφορά ότι οποιαδήποτε δυσμενής ε, ρύθμιση λόγω του γεγονότος ότι είχε τη δυσλεξία και δεν μπορούσε να αντιληφθεί πλήρως ε, την εφαρμογή όλων των κανονισμών οποιαδήποτε ε, δυσμενής μεταχείριση και ποινή η οποία του έχει επιβληθεί και ενδεχόμενα άλλα μέτρα να ζητούμε από τις αρμόδιες Ιρλανδικές αρχές να αρθούν διότι πρέπει πέραν του γεγονότος ότι ήρθε εδώ βεβαίως και είναι ένα παράδειγμα προς όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αγωνίζονται πρακτικά ο ίδιος να έχει και ένα αποτέλεσμα όχι μόνο να αλλάξει η συμπεριφορά η Ιρλανδία και οι άλλες χώρες για τον τρόπο επικοινωνίας, αλλά ο ίδιος να σταματήσει να υποβάλλεται στις δυσμενείς αυτές επιπτώσεις. Δηλαδή να αρθεί το πρόστιμο και οποιαδήποτε άλλη δυσμενής επίπτωση υπάρχει στη συγκεκριμένη περίπτωσή του. Ευχαριστώ. We'll take note of that and put... Το σημειώνουμε αυτό, θα το συμπεριλάβουμε και αυτό στην επιστολή και επίσης θα ε, καλέσουμε τις ε, αρχές να παρουσιάσουν γρήγορα αποτελέσματα. Καλό και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθήσει το θέμα αυτό στη συνέχεια και να βρισκόμαστε σε επαφή. Είμαι βέβαιη ότι μαζί θα μπορέσουμε να πετύχουμε κάποια αλλαγή. Σας ευχαριστώ κύριε Ντίερινγκ. Καλή επιστροφή στην Ιρλανδία, στο Πράσινο νησί. και μείνετε ήσυχος, ε, θα εξετάσουμε το θέμα αυτό στις επόμενες μέρες. Σας ευχαριστώ πολύ. Προχωράμε τώρα στην επόμενη αναφορά, 1003 σχετικά με τη μη εκπλήρωση εκ μέρου τη Πολωνία των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Δεν είναι παρόν ο αναφέρον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως είναι. Της δίνω το λόγο κατευθείαν. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η αναφορά αυτή σχετίζεται με τη μη εκπλήρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία εκ μέρους της Πολωνίας. Στην Πολωνία Είχαμε κάποιες εσωτερικές ε, επαφές. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βλέπει πολύ επικριτικά την ε, θέση του Πολωνού διαμεσολαβητή. Υποβλήθηκαν παράπονα σχετικά με τα νοικοκυριά, την φτώχεια στα νοικοκυριά ατόμων με αναπηρίες. Θέματα κοινωνικής ασφάλισης, αναφέρονται, αναφέρεται ότι δεν παρακολουθούνται επαρκώς τα επίπεδα φτώχειας. Και επίσης ότι δεν γίνονται αρκετές προσπάθειες ε, ώστε να διορθωθεί η κατάσταση. Δεν υπάρχουν ε, κέντρα αποκατάστασης. Και γενικά δεν ε, αντιμετωπίζονται τα προβλήματα των ανθρώπων με αναπηρίες. Ε, άλλωστε υπάρχει δυνατότητα χρήσης ε, των διορθωτικών ταμείων ε, για να υποστηριχθεί ανεξάρτητη διαβίωση. Τα στοιχεία που σχετίζονται με την κοινωνική ασφάλιση είναι θέματα στα οποία δεν μπορεί να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι ανησυχίες που αναφέρονται στην επιστολή βρίσκονται πέρα από τις αρμοδιότητες ε, της ε, Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Αλλά παρακολουθούμε την κατάσταση, κάθε χρόνο αναλαμβάνουμε δράσεις για <clears throat> την μείωση της φτώχειας και για να καλυφθούν οι ανάγκες ατόμων με, ειδικές, με αναπηρίες και να αντιμετωπιστεί ο αυξημένος κίνδυνος που έχουν τα άτομα με αναπηρίες σε σχέση με τα άλλα άτομα όσον αφορά τη φτώχεια. Ε, είναι θέμα με το οποίο ασχολείται η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας ε, και έχουμε επαφή με ένα δίκτυο εμπειρογνωμόνων στον τομέα αυτό. Έχουμε δημοσιεύσει πέρσι ε, μία έκθεση με μέτρα που μπορούν να ληφθούν για να βελτιωθεί η κοινωνική προστασία. ώστε ε, να επιτευθούν ε, καλύτερα οι στόχοι της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Όσον αφορά την ε, χρήση ευρωπαϊκών πόρων, αυτή είναι μια ανησυχία που επανέρχεται εδώ στην Επιτροπή. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε την υποστήριξη για την μετάβαση σε ανεξάρτητη διαβίωση. Κατά την ε, χρήση των πόρων θα πρέπει να ε, γίνεται σεβαστή και η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. και ε, αν υπάρχει συγκεκριμένος κανονισμός ε, σχετικά με την ε, χρήση των πόρων αυτών θα θέλαμε πολύ αναλυτικές πληροφορίες ώστε μαζί με τις εθνικές αρχές να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε την κατάσταση. Άλλωστε οι εθνικές αρχές είναι αυτές που έχουν την ευθύνη για την εφαρμογή. Πάντως με αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα ταμεία θα μπορέσουμε καλύτερα να απαντήσουμε στα θέματα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να αναφερθώ και σε μια επιστολή που λάβαμε από τις πολωνικές αρχές. όπου λένε ότι καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για εφαρμογή της σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Το Υπουργείο αναφέρει ότι υπάρχουν ε, ε, κοινέ αρμοδιότητες ανάμεσα στην Πολωνία και την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την πολιτική αυτή. Αναφέρονται στην αρχή της επικουρικότητας, ε, λένε ότι είναι θέμα των κρατών μελών να θεσπίσουν εθνικά μέτρα. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου καθώς και της σύμβασης στην οποία έχει προσχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την οποία έχει προσεπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει υποχρέωση να παρακολουθείται η κατάσταση σε όλα τα κράτη-μέλη. Στην περίπτωση αυτή νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να παρέμβει και γι' αυτό θα πρέπει να κλείσει αυτή η αναφορά και να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας. Αυτό θα κάνουμε λοιπόν. Σας ευχαριστώ θερμά. Προχωράμε στην επόμενη αναφορά. 11.32. Ε, έχει να κάνει με ε, την Jugend am Werk Steiermark GmbH ε, σχετικά με τη συμμετοχή ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας στην δημοκρατική ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι παρόν ο αναφέρον, ο κ. αν έχει το λόγο για πέντε λεπτά. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σήμερα εκπροσωπώ τα άτομα με ε, πολύπλοκες ε, αναπηρίες ε, και προβλήματα ψυχικής υγείας και αναφορά μου έχει να κάνει με τα έτη 2015-2016 και τις ε, εκδηλώσεις σε διάφορα κράτη-μέλη όπου ε, κλήθηκαν ε, άτομα με αναπηρίες να διατυπώσουν τις προτάσεις τους για καλύτερη συμμετοχή τους ε, στη δημοκρατική ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, το ότι βρίσκομαι εγώ εδώ σήμερα, αλλά κανένας από αυτούς τους ανθρώπους, ε, σημαίνει ότι ο στόχος δεν είχε επιτευχθεί καθόλου. Και άτομα με πολύπλοκες αναπηρίες δεν είναι σε θέση μέσα σε πέντε λεπτά να παρουσιάσουν το πρόβλημά τους εδώ στην Επιτροπή τους. Και για πολλά από τα άτομα αυτά δεν είναι καν δυνατόν να παρακολουθήσουν τη συζήτηση που διεξάγουμε εδώ πέρα, ούτε με βοήθεια των πολλών τεχνικών δυνατοτήτων που προσφέρονται εδώ πέρα. Τι χρειάζονται λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να συμμετάσχουν στην ε, δημοκρατική ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε πολλές ε, συζητήσεις, ε, εργαστήρια κατά τη διάρκεια του προγράμματος ε, που πραγματοποιήσαμε πάνω στο θέμα αυτό. Σε όλες τις χώρες ένα θέμα τονιζόταν. Ανάγκη για σεβασμό. Σεβασμός και ισότητα. Και τι χρειάζεται. Χρειάζεται χρόνος να ακούσει κανείς, να καταλάβει τα προβλήματα των ανθρώπων αυτών και να δώσουν εξηγήσει. Μάλιστα, αυτά, ε, ο χρόνος αυτός χρειάζεται και από τις δύο πλευρές. Και μέρος αυτού είναι η βούληση. Αυτό ε, σημαίνει η ενεργός συμμετοχή δεν ε, σημαίνει το ίδιο που σημαίνει για όλους εδώ ε, το να μπορούμε να διαβάσουμε, να γράψουμε, να παρακολουθήσουμε. Σήμερα υπάρχουν ε, τεχνικές δυνατότητες οι οποίες προσφέρουν πολλές δυνατότητες αλλά υπάρχουν λήψεις όσον αφορά τα πρότυπα και την εφαρμογή τους. Χρειαζόμαστε λοιπόν ε, όχι μόνο πιο ε, απλή διατύπωση, πιο καλή αναγνωσιμότητα, αλλά και πιο καλή ε, διατύπωση, χρήση της γλώσσας και χρήση εικόνων. Άτομα με με προβλήματα εκμάθησης και πολύπλοκες ε, αναπηρίες ε, θέλουν μεταξύ άλλων ε, και να εργαστούν. Οι άνθρωποι αυτοί δεν θέλουν να είναι εξαρτημένοι από το κοινωνικό κράτος, θέλουν να συμβάλλουν και εκείνοι. Και γι' αυτό ζητούν προσφορά εκπαίδευσης προσαρμοσμένης στα μέτρα τους. Θέλουν να μπορούν να, να βγάλουν μόνο τους τα χρήματά τους ε, και να μπορούν να συμβάλλουν στην κοινωνία και να πάρουν σύνταξη. Ο σεβασμός ε, σημαίνει για τους ανθρώπους αυτούς ε, να μπορούν να συμμετάσχουν στη λήψη αποφάσεων και ιδιαίτερα αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή τους. Αυτό έχει να κάνει και με τον δημόσιο και με τον ιδιωτικό βίο. Και στα δύο αυτά πλαίσια θα πρέπει να εφαρμοστούν οι βασικές αρχές. θέλουν εξάλληψη των εμποδίων ε, στην επικοινωνία. Πέρα από αυτό όμως αναφέρθηκε και η κοινωνική και πολιτική εκπροσώπηση καθώς και η δυνατότητα αυτοεκπροσώπησης. Τέλος, ε, θα ήθελα να πω ότι εάν ε, η ένταξη γίνει πραγματική συμμετοχή των ε, ανθρώπων αυτών. Εάν δεν θέλουμε απλά να παραμείνει λόγια στο χαρτί, θα πρέπει να δίνουμε τις προσπάθειές μας. Ήδη έχουν γίνει πολλά. Ωστόσο, στο πλαίσιο του προγραμματός μας ε, φαίνεται ότι τα μέτρα ε, δεν ε, φτάνουν πάντα, δεν ωφελούν πάντα τους ανθρώπους για τους οποίους ε, προορίζονται και αυτό το έδειξε και η προηγούμενη υπόθεση που ακούσαμε από την Ιρλανδία. Γι' αυτό καλώ τους πολιτικούς εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εντείνουν τις προσπάθειες σύμφωνα και με την αναφορά μας, ώστε να υπάρχει ίση συμμετοχή ατόμων ε, με προβλήματα εκμάθησης και πολύπλοκες ε, αναπηρίες, ε, ώστε να ωφεληθούν τα άτομα αυτά από τα σχετικά μέτρα. Σας ευχαριστώ. Να τονίσω ότι δεν βλέπετε μεν πολλούς στην αίθουσα. Παρ' όλα αυτά η συνάντηση αυτή είναι διαθέσιμη μέσα από το δίκτυο και γνωρίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι και αρμόδιοι υπάλληλοι οι οποίοι παρακολουθούν ε, γιατί οφείλουν να είναι σε μια διαφορετική αίθουσα. Αυτό το βλέπω στο τηλέφωνο μου. Κάνουν ε, αναφορές σε αυτά τα οποία κάνουν, συμμετέχουν, σημειώνουν και ευχαριστούν. Αυτό σημαίνει ότι σας άκουσαν χιλιάδες ε, ακροατές κατά τη διάρκεια της παρέμβασής σας. Είναι καλό να το γνωρίζετε. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Θα ξεκινώντας ευχαριστώντας τον αναφέροντα που εξέφρασε με ξεκάθαρο τρόπο την κατάσταση σχετικά με τη συμμετοχή των προσώπων των ατόμων που έχουν προβλήματα στον τομέα της ε, με διανοητικές μορφές αναπηρίας και αντίστοιχες τέτοιες περιπτώσεις. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να επιτραπεί η συμμετοχή τους στις πολιτικές διαδικασίες ισότιμα και στην εκπαίδευση, στην απασχόληση που υπογραμμίσατε. Τίθεται φυσικά το θέμα έντονα της πολιτικής συμμετοχής, της, της συμμετοχής στα πολιτικά τεκτενόμενα. Είναι σημαντικό να υπογραμμίσει κανείς ότι η αναφορά αυτή προκλήθηκε από ένα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, είμαστε ικανοποιημένοι γιατί βλέπουμε ότι η χρηματοδότηση αυτή, το πρόγραμμα αυτό, ε, βοηθά στο να συνειδητοποιηθεί το πρόβλημα και η πρόκληση και ίσως και με μεγαλύτερη ταχύτητα. Έχουμε ένα εξαιρετικό μέσο, τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ανθρώπων με Αναπηρίες, Υπάρχουν συγκεκριμένες βασικές αρχές οι οποίες μας επιτρέπουν να βρούμε λύσεις με βάση τα άρθρα 9, 21 και 30 για τα θέματα της συμμετοχής στις πολιτικές διαδικασίες και άλλα άρθρα σχετικά με την εργασία κτλ. Πάντως αυτό το οποίο έχει σημασία να πω είναι ότι τα άρθρα αυτά δεν είναι κάτι το τυπικό, το ονομαστικό απλά αλλά το θέμα είναι να προσπαθήσουμε να τα μετατρέψουμε σε κάτι το πραγματικό. Θα μπορούσα να σας δώσω κάποια παραδείγματα σχετικά με την πρόσβαση στην ενημέρωση. Όταν διοργανώνουμε κάποιες εκδηλώσεις βάζουμε στην ημερήσια διάταξη θέματα τα οποία ανησυχούν τους πολίτες. Επιλέγουμε θέματα σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών Όλα αυτά καθίστανται διαθέσιμα σε μορφή προσβάσιμη. Όπως και σήμερα υπάρχει η διαδικασία speech to text, δηλαδή από την ομιλία σε γραπτό κείμενο κτλ. Πάντως, σε σχέση με τα θέματα της ενημέρωσης, να πω ότι παίρνουμε και κάποιες, κάποια μέτρα τα οποία έχουν σαν στόχο να ενημερώσουν σωστά για τις εξελίξεις σε νομικό επίπεδο. Σαν παράδειγμα, εμείς κάνουμε την πρόσβαση στις ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο προσβάσιμες. Συζητάμε το θέμα της Ευρωπαϊκής Πράξης για την, για την προσβασιμότητα για να καταστήσουμε προσβάσιμες υπηρεσίες και προϊόντα που στο παρελθόν δεν ήσαν προσβάσιμα. Μόνον έτσι θα μπορέσουμε να δώσουμε την δυνατότητα στους πολίτες με αναπηρίες να μπορέσουν να κάνουν και επιλογές και να πάρουν τις σωστές αποφάσεις. Ταυτόχρονα στις αποφάσεις που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει και το θέμα του κατανοητού των ευρωπαϊκών εγγράφων και αποφάσεων. Στον τομέα της εκπαίδευσης δεν ξέρω αν ήσασταν εδώ από το πρωί αλλά συνεργαζόμαστε με την υπηρεσία, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εκπαίδευσης χωρίς αποκλισμούς και με τις αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών μελών. Θα μπορούσα να σας δώσω και περισσότερα παραδείγματα <clears throat> Σαν παράδειγμα συμπεριλαμβάνουμε στο Erasmus Plus φοιτητέ οι οποίοι έχουν δυσκολίες πρόσβασης και οι οποίοι είναι σε θέση να διαπιστώσουν τις συνθήκες ένταξής τους στο πρόγραμμα αυτό. Κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι όταν προσπαθούμε να προκαλέσουμε τη συνειδητοποίηση και του θέματος και την κατανόηση του, θέματος, του θέματος έμεσα. Αυτή είναι μια διαδικασία που βοηθά να συνειδητοποιήσει ακριβώς ο κόσμος και το βάθος του προβλήματος. Αλλά πάντως όπως είπα ε, η εφαρμογή της σύμβασης ε, είναι κατανεμημένη αρμοδιότητα αφορά και στα κράτη-μέλη και σε εμάς. Εμείς συλλέγουμε στοιχεία, συλλέγουμε δεδομένα, συλλέγουμε δείκτες, αλλά τελικά κάθε εμπλεκόμενος οφείλει να καταθέσει μια έκθεση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο φέρει πέρα στις υποχρεώσεις του ιδιαίτερα σε τομείς όπου μπορεί να είναι εκτός ε, του κοινοτικού πλαισίου. Πάντως αναφέρθηκα και σε οδηγίες όπως η προσβασιμότητα της, των ιστοσελίδων των ευρωπαϊκών οργάνων είναι πρακτικά δείγματα θα έλεγα της προσπάθειάς μας η συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Πράξη για την Προσβασιμότητα οδηγούν ακριβώς τα στάνταρτ τα οποία συνοδεύουν τις αποφάσεις που λαμβάνουμε σε νομοθετικό επίπεδο καθιστώντας για όλες τις κατηγορίες αναπηρίας προσβάσιμα στοιχεία ενημέρωσης και πληροφόρησης μεταξύ των οποίων και θέματα που άπτονται των διανοητικών αναπηριών. Δεν ξέρω ποιος θα ήθελε το λόγο, ο κύριος Μαριάς ή η κυρία Ιστάρας. Σας ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα των αναφερόντων. Πράγματι η συγκεκριμένη αναφορά θα έλεγα συμπυκνώνει την μεγάλη συζήτηση της αναπηρίας όπως επίσης και της προσβασιμότητας στην Ευρώπη της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς της υγείας, της κατοικίας κτλ. Όπως είπε και η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εμείς εργαζόμαστε γύρω από το θέμα της Ευρωπαϊκής Πράξης για την Προσβασιμότητα και τα πολλαπλά προγράμματα που θα προέρχουν από αυτή. Θα ξεκινήσουμε ε, σύντομα, θα ξεκινήσουμε έλεγα σύντομα την διαδικασία του τριμερούς διαλόγου εμείς έχουμε φυσικά τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών που είναι η βάση ε, για τις ε, ε, προσπάθειές μας και εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πλαίσια του δικτύου μας και σε συνεργασία με τη διαμεσολαβήτρια ενημερώνουμε όλες τις χώρες μέλη όπως και την Αυστρία για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζουν την σύμβαση αυτή. Λέγεται ότι θα πρέπει να επιβλέπεται η εφαρμογή της ε, συγκεκριμένη σύμβασης και γι' αυτό μπορούμε να κρίνουμε το τι ακριβώς συμβαίνει σε όλες τις χώρες μέλη. θα εξαρτηθεί η προσπάθεια αυτή που κάνουμε από τις ε, ενέργειες τις οποίες κάνει το network που έχουμε σε σχέση με τα θέματα εφαρμογής και θέλει να είναι θέλουν να είναι ενημερωμένα τα Ηνωμένα Έθνη για τον τρόπο με τον οποίο εμείς εφαρμόζουμε τις προτάσεις τους. Αναφέρθηκε σε αυτό η Μακολάδα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αν δεν υπάρχει σωστή εφαρμογή να δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να διορθώσουμε την κατάσταση. Το θέμα δεν είναι μία περίπτωση κάθε φορά, το θέμα είναι γενικό σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει η Επιτροπή. Και από αυτή την αναφορά να αναδεικνύονται τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ειδικέ ανάγκες. Ε, το βασικό είναι η προσβασιμότητα και νομίζω ότι προέχει να βρούμε τον τρόπο, το σωστό τρόπο εφαρμογής της ε, ε, Διεθνούς ε, Σύμβασης του ΟΗΕ. Ο στόχος ε, είναι να βοηθήσουμε. Αυτό είναι το βασικό. Έχουμε πάρα πολλές αναφορές για τα ζητήματα αυτά. Θεωρώ σημαντική την σημερινή ημέρα έτσι όπως εξελίσσεται με τις παρεμβάσεις και το workshop που είχαμε ε, και φυσικά χωρίς τη συνεργασία της Κομισιόν και των κρατών μελών δεν μπορεί να προχωρήσει το όλο εγχείρημα. <clears throat> Όμως δεν θα πρέπει οι δυσκολίες που υπάρχουν να αποτελούν άλοθη για τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη έχουν υποχρεώσεις. Θα πρέπει να υπάρξει σωστή εφαρμογή της ε, Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ. Και φυσικά θα πρέπει να φέρουν αποτελέσματα, να δώσουν ε, πραγματικά οδηγίες, να πάρουν μέτρα. Διότι τα άτομα με αναπηρίες δεν μπορούν να περιμένουν πότε κάποιο κράτος μέλος θα δεήσει, θα αποφασίσει να συμμορφωθεί. Επομένως, ε, μαζί με τη συνεργασία πρέπει να υπάρξει και η πίεση, η αποφασιστική πίεση στα κράτη ούτως ώστε να συμπορφωθούν. Νομίζω ότι προφανώς θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά, να ασκήσουμε την μέγιστη δυνατή πίεση προς τις αρχές της Αυστρίας, αλλά να είναι και ένα μήνυμα προς τα υπόλοιπα κράτη-μέλη ότι εμείς εδώ ως Επιτροπή και ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε αποφασισμένοι να στηρίξουμε τα άτομα με αναπηρίες διότι δεν μπορούν να έχουν δυσμενή μεταχείριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ όλους. Καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ τους αναφέροντες, διότι η αναφορά σας ήταν πολύ επίκαιρη ε, το 2016 που έγινε. Μετά το 2016 έχουν συμβεί πολλά. Ακούσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τους συναδέλφους ε, ε, και άλλους στη διάρκεια της ακρόασης. Ε, υπάρχει μία δέσμευση που δεν υπήρχε το 2016 και η πράξη της προσβασιμότητας που εκπονούμε τώρα, ε, η οδηγία για την πρόσβαση στο διαδίκτυο που ε, εξετάζουμε τώρα, όλα αυτά είναι θέματα προσβασιμότητας στη διάρκεια των εκδηλώσεων, πιο εύκολη γλώσσα, νέε τεχνολογίε, όλα έχουν ληφθεί υπόψη με τρόπο που δεν συνέβαινε όταν ε, υποβάλλετε την αναφορά σας. Μια μεγάλη νίκη για σας. Καταφέρατε πολλά. Ε, μπορείτε να επιστρέψετε και να πείτε στους φίλους και στου συναδέλφους σα ότι ήταν μια πάρα πολύ σημαντική συνεισφορά σας στην όλη διαδικασία και από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ε, τώρα πρέπει να τη συνοδεύσουμε. Η κατάσταση έχει αλλάξει γιατί η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών ε, πλέον ε, έχει κυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη μεγάλη πλειοψηφία των κρατών μελών. Όπως είπε και ο κύριος Μαριάς, πλέον πρόκειται για μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Η πρόκληση είναι πώς ε, θα την εφαρμόσουμε. Και ε, σε αυτό βασιζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να παρακολουθήσει τη διαδικασία και να ε, μας αναφέρει αν υπάρχουν ε, παρατυπίες ε, ε, σε κάποιο από τα κράτη-μέλη. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν, αλλά για πάνε ενδεχόμενο βασιζόμαστε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακούσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η υπόθεση είναι ξεκάθαρη, βοηθήσατε ιδιαίτερα στην όλη διαδικασία και τα θέματα που θίξατε ελήφθησαν υπόψη και στη διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, ε, και εμείς από πλευράς Επιτροπής Αναφορών ε, κοινοποίησαμε την Επιτροπή Απασχόλησης για το θέμα και γι' αυτό ακριβώς θεωρώ ότι είναι και η στιγμή να την κλείσουμε. Διότι η συμβολή σας ήταν ε, πολύ σημαντική, τη λάβαμε υπόψη, βλέπω ότι γνέφετε, συμφωνείτε κι εσείς. Νομίζω λοιπόν ότι μπορείτε να συνεχίσετε πλέον τη ζωή σας και να ασχοληθείτε με κάτι άλλο, να επενδύσετε την ενέργειά σας κάπου αλλού. Ε, που θα χρειάζεται και τις, ικανότητες, σας, τις ικανότητές σας. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι τομεί και στην Αυστρία. Σας ευχαριστούμε πολύ και θα κλείσουμε την αναφορά και περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχή συνεργασία για τη διαδικασία εφαρμογής. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα περνάμε στην επόμενη αναφορά, που είναι η αναφορά 0857 της κυρίας Ρωμίνα Φρασάνη για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα στη Ρουμανία. Έχουμε εδώ την αναφέρουσα. Σας δίνουμε το λόγο για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω. Φέτος είναι 10 χρόνια από τότε που εντάχθηκε η Ρουμανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει, ότι υποστηρίζει πλήρως την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα άτομα με αναπηρία και πολλοί επικεντρώνονται στην εφαρμογή και την προστασία αυτής της ε, σύμβασης. Είναι λοιπόν επονίδιστο το γεγονό ότι βλέπουμε ότι μετά από 10 χρόνια εφαρμογή ε, ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει εφαρμόσει η Ρουμανία και έχει αγνοήσει πλήρω τι ευθύνε τη βάση τη σύμβαση. Η σύμβαση μεταξύ άλλων ζητά πλήρη ε, πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες και πρόσβαση σε δημόσιες κοινωνίες. Εγώ είμαι σήμερα για να ζητήσω ε, από την Επιτροπή να αναλάβει δράση για την προστασία των πολιτών. Η Ρωμία ε, δεν μπορεί να απολαμβάνει μόνο τα ωφέλη τη ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να αγνοεί τι υποχρεώσει. Δεν είναι πλέον καινούριο μέλο και δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αυτό ω αιτιολογία. Ο πληθυσμό είναι πάνω από 20 εκατομμύρια και είναι προφανώ ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση υπηρεσιών τρένου. Ε, οι δημόσιες συγκοινωνίες είναι πολύ σημαντικές για τη Ρουμανία. Το σιδηροδρομικό δίκτυο επιτρέπει ε, μεταφορά για την εργασία, την εκπαίδευση και τα ταξίδια. Επομένως είναι πάρα πολύ ανησυχητικό το γεγονός ότι στην όλη χώρα δεν υπάρχει προσβάσιμο τρένο και θα μπορούσατε να πάτε και στο μεγαλύτερο τρένο στη Ρουμανία, στη, ε, στο Βουκουρέστι, δεν υπάρχει πρόβλεψη για τα άτομα με αναπηρία. Η Ρουμανία ε, υποσχέθηκε να προστατεύσει τα δικαιώματα των πολιτών, αλλά φαίνεται να λησμονεί αυτούς που έχουν κάποιες αναπηρίες. Ε, και σε αυτή την περίπτωση είναι άτομα τα οποία χρειάζονται προστασία και δεν ξέρω γιατί δεν θεωρούνται τόσο σημαντικά. Ε, επειδή ακριβώ δεν εκμεταλλεύεται το σύστημα, στερεί τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία να έχουν ίση πρόσβαση σε αυτέ τι υπηρεσίε όπω όλοι οι υπόλοιποι. Για να ταξιδέψει κάποιο με τρένο στη Ρουμανία, θα πρέπει να περάσει από μια μακροβόρα και πολύ άδικη διαδικασία, για να είμαι ειλικρινής πρέπει να έρθουν σε επαφή με τον ε, σταθμάρχη απευθείας, γραπτός, τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν, για να ζητήσουν άδεια για να ταξιδέψουν και η άδεια από εκεί και πέρα επαφίζει στη διακριτική ευχαίρεια του διευθυντή. Ακόμα και το εγκρίνει δεν σημαίνει ότι κάποιο θα μπορέσει να ταξιδέψει. Για του χρήστε αναπηρικού αμαξιδίου, για παράδειγμα, το θέμα τη φυσική πρόσβαση είναι πρόβλημα. Όλα τα τρένα έχουν στενέ εισόδου με τρία πολύ ψηλά σκαλοπάτια. Και όταν ρώτησα, μου είπαν ότι θα μπορούσε να γίνει κάποια ρύθμιση για να με σηκώσουν, αλλά θα πρέπει να περάσω όλο το ταξίδι ε, μέσα ε, μπροστά στην πόρτα του τρένου. Επίση, να σα πω ότι τα ταξίδια στο Ρουμανία διαρκούν ε, πάνω από 8 ώρε που σημαίνει ότι θα κάτσω 8 ώρε μπροστά στην πόρτα. Ε, εάν κάποιο ε, ο οποίο δεν είχε κάποια αναπηρία θα ήταν υποχρεωμένο να ταξιδέψει έτσι, θα είχε δημιουργηθεί μεγάλη αναστάτητα. Τα τρένα δεν προσφέρουν καμία πρόσβαση. Αυτοί που έχουν προβλήματα κινητικότητα δεν μπορούν να περάσουν από την είσοδο και να πάνε στην, στο βαγόνι που υπάρχουν ε, θέσεις. Ε, και επίσης δεν υπάρχει πρόσβαση ε, σε τουαλέτα. Εκτός και αν είσαι κάποιος ο οποίος έχει πλήρη υγεία, το ταξίδι είναι πάρα πολύ δύσκολο και σχεδόν αδύνατο για άτομα σαν εμένα. Ως πολίτης της Ευρώπης θυμάμαι μια άλλη εποχή της ιστορίας που οι τέλειοι άνθρωποι ήταν οι ευνοούμενοι και οι υπόλοιποι δεν, έτυχαν, δεν τύχαναν του ίδιου συμβασμού. Ήρθα εδώ για να μιλήσω για το σιδηροδρομικό σύστημα στη Ρουμανία, αλλά όπω είδαμε το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό. Τα άτομα με αναπηρία δεν έχουν βασικά δικαιώματα σε παιδεία, απασχόληση, ακόμα και τη δυνατότητα για κοινωνική ζωή. Κάποιοι δεν έχουν καν την πολυτέλεια να βγουν από το σπίτι του. Και ε, πολύ συχνά στα κανάλια τηλεοράσεων βλέπουμε ανθρώπου που δεν έχουν βγει ποτέ, δεν έχουν πάρει καθαρό αέρα ή κάποιο ηλικιωμένο πατέρα που χρειάζεται να κουβαλάει το παιδί του πάνω κάτω σε 50 σκαλοπάτια για να μπορεί να έχει πρόσβαση στην εκπαίδευση και να φτάνει στο σχολείο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπακούν σε όλους τους κανόνες και όχι επιλεκτικά σε κάποιους. Η Ρουμανία θα πρέπει να κάνει κάτι και από αυτά που έχει δεσμευτεί να κάνει. Υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα που έχει υποσχεθεί η ρουμανική κυβέρνηση για να παρέχει υπηρεσία σε άτομα με αναπηρία, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί κανένα από αυτά. Είναι πονίδιστο εν έτη 2017 η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην μπορεί να είναι περήφανη για όσα έχουν επιτύχει τα κράτη-μέλη της. Ακόμα και κάτι πολύ απλό όπως το να ακούν τους κανόνες. Για τον υπόλοιπο κόσμο φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια περιοχή με ίσα δικαιώματα και ευκαιρίε. Αλλά πόρα απέχουμε από αυτή την κατάσταση. Η Ρουμανία πρέπει να τιμωρηθεί ε, γιατί δεν αναλαμβάνει δράση. Όχι μόνο δεν αρνείται πρόσβαση, αλλά και σε Ευρωπαίου πολίτε ε, που δεν μπορούν να ταξιδέψουν και να θαυμάσουν τι ομορφιέ τη Ρουμανία δεν προσφέρεται η ίδια ευκαιρία. Θα πρέπει λοιπόν να τηρηθεί η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών. Είναι σκανδαλώδες το ότι δεν εφαρμόζεται. Το θέμα της πρόσβασης σε μεταφορές θα πρέπει ε, να ληφθεί υπόψη και όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν και να ζουν φυσιολογική ζωή στα σύνορα. Τα άτομα με αναπηρία ήδη αντιμετωπίζουν πολύ σημαντικές προκλήσεις στη ζωή όπως είδαμε. Θα πρέπει τουλάχιστον να εξασφαλίσουμε ότι θα ε, έχουν τη στήριξη της κυβέρνησής τους και η κυβέρνηση θα προστατεύσει τα δικαιώματά τους. Σήμερα θα ήθελα να σας ζητήσω να θυμηθείτε ότι ναι μεν τα άτομα με αναπηρία είναι μειονότητα, ο, κανέ, ο καθένας, ακόμα και ο καθένας από εσά θα μπορούσε να γίνει κάλλιστα άτομα με αναπηρία και να νίκει στην ομάδα λόγω μιας ασθένειας. Θα ήθελα να ολοκληρώσω να σας ευχαριστήσω για την ε, βοήθειά σα και όλους εκείνους που συμμετέχουν στη στήριξη των ατόμων με αναπηρία και να σας ευχαριστήσω και για τη δυνατότητα να συμμετέχω στη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, ε, προσπαθήσατε να καλέσετε του ευρωβουλευτής, ευρωβουλευτές και άλλους να ταξιδέψουν μαζί σας στο τρένο. Εγώ το έκανα αυτό στη Σουηδία. Ε, να γίνετε ακτιβίστρια εάν δεν μπορέσετε να τους ε, κινητοποιήσετε. Τουλάχιστον έχετε δύο υποστηριχτές μπροστά σας. Εμείς θα έρθουμε. Ε, προσπάθησα να έρθω σε επαφή μαζί τους ε, πριν ε, έρθω εδώ σήμερα. Ε, ε προσπάθησα να έρθω σε επαφή με μέλη δύο διαφορετικών κομμάτων και με αγνώρισαν τελείως. Ε, αυτό είναι ακόμα πιο ε, ε, κακό. Πάντως έχετε υποστηριχτές από την Ισπανία, τη Σουηδία, την Ελλάδα. Θα πάμε όλοι μαζί. Και είμαι βέβαιη ότι θα συμμετάσχουν και άλλοι, διότι αυτό είναι σκανδαλώδες, τελεία. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζω να μπορέσουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας στο θέμα αυτό. Ναι, φυσικά και η Ρουμανία στηρίζει τις προσπάθειες ε, πολιτών ε, με αναπηρίες ε, και καταλαβαίνουμε απολύτως τις δυσκολίες της αναφέρουσας κατά την χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς και ιδιαίτερα στη Ρουμανία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών, όπως είναι το δικαίωμα μη διάκρισης και Σύμφωνα και με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα άτομα με αναπηρίες, ε, έχει αναλάβει μια σειρά δράσεων ε, για άτομα με αναπηρίες ε, ή με μειωμένη κινητικότητα θα ήθελα να πω λίγα λόγια σχετικά με το τι έχουμε κάνει για τα δικαιώματα των επιβατών. Για άτομα με περιορισμένη κινητικότητα και με αναπηρίες. Κάτι που σχετίζεται και με τις ε, τεχνικές ε, ε, προδιαγραφές για τη διαλειτουργικότητα. Και ίσως ο συνάδελφος να θέλει να προσθέσει κάτι για την Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας. Αυτή τη στιγμή έχουμε τον κανονισμό 1375 του 2007 για τα δικαιώματα των επιβατών που ταξιδεύουν με τρένο. Ο κανονισμός αυτός ήδη περιέχει κάποιες διατάξεις για άτομα με μειωμένη κινητικότητα ή με αναπηρίες, αλλά πιο πολύ έχει να κάνει με την παροχή πρόσθετης βοήθειας ε, παρά με την ε, προσβασιμότητα των τρένων. Δυστυχώς ε, αυτή τη στιγμή υπάρχει δυνατότητα για τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν μια σειρά από παρεκκλήσεις για τις εγχώριες μεταφορές και η Ρουμανία έχει εκμεταλλευτεί πολύ αυτή τη δυνατότητα. Έχει παρέκκληση για όλα τα υποχρεωτικά άρθρα του κανονισμού που σχετίζονται με τις ε, υπηρεσίες που πρέπει να παρέχονται σε άτομα με αναπηρίες ή με περιορισμένη κινητικότητα στο τρένο και στους σταθμούς. Αυτό σημαίνει ότι τα περισσότερα από αυτά τα άρθρα πέρα από το άρθρο για τις μη διακρίσεις και το άρθρο που σχετίζεται με τις πληροφορίες που θα πρέπει να παρέχονται σχετικά με την προσβασιμότητα του συστήματος ε, σιδηροδρομικών μεταφορών ε, για όλα τα υπόλοιπα άρθρα λοιπόν υπάρχει παρέκκληση στη Ρουμανία. Θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις ε, τεχνικές προδιαγραφές για τη διαλειτουργικότητα για τα άτομα με ε, μειωμένη κινητικότητα ή με ε, αναπηρίες, το οποίο σημαίνει ότι το τροχαίο υλικό και η υποδομή των σιδηροδρόμων, δηλαδή και τα βαγόνια και οι σταθμοί και το περιβάλλον τους θα πρέπει βαθμιαία να γίνουν προσβάσιμα. Το οποίο σημαίνει ότι κάθε φορά που οικοδομείται νέο σταθμό ή που ε, τίθενται σε λειτουργία νέα τρένα, αυτά θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις προδιαγραφές. Ε, βαθμιαία όμως σημαίνει ότι ε, όσον αφορά το υπάρχον τροχαίο υλικό και τους υπάρχοντες σταθμούς δεν χρειάζεται να γίνει τίποτα εκτός εάν υπάρξει αναβάθμιση ή ανακαίνιση και επίσης ε, δεν ε, ισχύουν ε, προθεσμίες για να γίνουν προσβάσιμα και υπάρχει το Συμβούλιο το οποίο επανεξετάζει την υπόθεση. Η Ρουμανία συμμετέχει σε αυτή τη Συμβουλευτική Επιτροπή, οπότε γνωρίζει ακριβώς τι διακυβεύεται όσον αφορά τον ε, κανονισμό 1371 του 2007 για τα δικαιώματα των επιβατών ε, και τις υποχρεώσεις ε, στις 20 Σεπτεμβρίου, τώρα μόλις δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει οθετήσει πρόταση για την αναθεώρηση του κανονισμού αυτού. Και η πρόταση αυτή περιέχει μια σειρά από για να επιτρέψει πιο εύκολα σε άτομα με αναπηρίες ή με περιορισμένη κινητικότητα να χρησιμοποιούν σιδηροδρομικές μεταφορές. Η πιο σημαντική ε, τροποποίηση είναι ότι θα μειώσουμε τις ε, παρεκκλήσεις ώστε ιδιαίτερα το κεφάλαιο 5 που περιέχει τα δικαιώματα των ε, ατόμων με αναπηρίες ή περιορισμένη κινητικότητα θα γίνει υποχρεωτικό στην πρόταση αυτή. Οι παρεκκλήσεις θα πρέπει να μειωθούν γενικά και Ειδικά το κεφάλαιο 5 για τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες ε, θα γίνει υποχρεωτικό για όλες ε, τις ε, υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών. Και όχι μόνο αυτά, πέρα από το θέμα των παρεκκλήσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης προτείνει βελτίωση της πληροφόρησης. Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται θα πρέπει να παρέχονται σε τρόπο, με τρόπο προσβάσιμο για άτομα με όλων των ειδών της αναπηρίας, όχι μόνο για τυφλούς και κοφούς. Επίσης, ε, προτείνουμε πρόσωπα που δεν μπορούν για λόγους προσβασιμότητας να αγοράσουν εισιτήριο στον σταθμό, επειδή ε, δεν υπήρχε προσβάσιμος τρόπος αγοράς του εισιτηρίου, να μπορούν να αγοράσουν το τρένο στο τρένο χωρίς επιπλέον χρέωση. Επίσης ε, προτείνουμε να παρέχετε βοήθεια ανα πάσα στιγμή κατά τη λειτουργία του τρένου και σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό και θα ήθελα να αναφερθώ στο, στο διάστημα κοινοποίησης που αναφέρατε. Ε, ο ισχύων κανονισμός ε, απαιτεί από τα άτομα με αναπηρίες ε, να κοινοποιήσουν 48 ώρες εκ των προτέρων τις ανάγκες τους. Εάν όμως γίνουν υποχρεωτικές αυτές οι διατάξεις. Αυτό θα ισχύει και για την Ρουμανία, το οποίο σημαίνει ότι αν ε, η επιχείρηση σας ζητάει ε, κοινοποίηση πριν, δύο εβδομάδες πριν, το οποίο είναι εξωφρενικό σύμφωνα απολύτως, τότε θα μπορέσετε να προσφύγετε ε, στην Εθνική Αρχή Επιβολής του Νόμου. Και όσον αφορά την, ε, τον εξοπλισμό ε, κινητικότητας εάν χαθεί θα πρέπει να καλύπτεται το κόστος και επίσης εάν παρέχεται προσωρινά άλλο είδος εξοπλισμού θα πρέπει να είναι αντίστοιχο με αυτό που χρησιμοποιείται. Επίσης, ε, εισάγουμε υποχρεωτική κατάρτιση του προσωπικού που παρέχει τη βοήθεια στα τρένα και στους σταθμούς. Αυτό δεν είναι υποχρεωτικό αυτή τη στιγμή σύμφωνα με τον κανονισμό, αν ε, και είναι ε, σύμφωνα με την ομοθεσία για άλλα είδη μεταφορών. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις λοιπόν θα πρέπει να καταρτίζουν το προσωπικό τους ώστε να μπορούν να παρέχουν βοήθεια ε, κατάλληλη για, που να καλύπτει τις ανάγκες ε, των ε, ατόμων με αναπηρίες. Και τέλος, βελτιώνουμε και την διαδικασία προσφυγής. και για άλλους φορείς πέρα από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και θα υπάρχει δυνατότητα να ε, ε, υποβάλει κανείς ε, τα παραπονά του κατευθείαν στο σταθμό. Αυτά λοιπόν τα νέα μέτρα που υιοθετήθηκαν πριν τρεις εβδομάδες. Είχαμε δύο συναντήσεις στο Συμβούλιο, άλλες δύο θα πραγματοποιηθούν εντός του μήνα. Η Εστονική Προεδρία πιέζει για να προχωρήσει το θέμα αυτό και θα αγωνιστούμε ώστε να παραμείνουν αυτές οι πολύ βασικές διατάξεις στον κανονισμό. Σας ευχαριστώ πολύ. να προσθέσω κάποια πράγματα. Η συνάδελφος μου έδωσε μια πολύ πλήρη ε, περιγραφή της ε, κατάστασης όσον αφορά την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ θα ήθελα να τονίσω ότι η Ρουμανία έχει επικυρώσει τη σύμβαση το 2011. Ε, ε, υπέγραψε το προαιρετικό πρωτόκολλο, δεν έχει επικυρωθεί όμως, το οποίο σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να αποστέλλονται ε, κοινοποιήσεις στην Επιτροπή, αλλά θα ήθελα να καλέσω τους αναφέροντες να έρθουν σε επαφή με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για τα θέματα αυτά. Η Ρουμανία θα πρέπει να υποβάλει δική της έκθεση και η κοινωνία των πολιτών μπορεί να αποστέλει εναλλακτικές εκθέσεις ε, που να περιγράφουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζεται. Η Επιτροπή αυτή εξετάζει πολύ ε, σοβαρά όλες τις αναφορές και είναι σημαντικό να διαδίδεται τις πληροφορίες αυτές, διότι ε, είναι σαφές όχι όσον αφορά μόνο την τις ε, σιδηρομικές ε, επιχειρήσεις για οποιαδήποτε υπηρεσία παρέχεται στο ε, κοινό από δημόσιο ιδιωτικό φορέα για τις υπηρεσίε αυτές η Ρουμανία έχει πρόσθετες υποχρεώσεις ε, σύμφωνα με την ε, σύμβαση όπως ε, επίσης και σύμφωνα με το άρθρο 20 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ανθρώπων με Αναπηρίες. Να σας διαβεβαιώσω λοιπόν ότι οι εμπειρίες που σας περιέγραψε η συνάδελφος σχετικά με τις παρεκκλήσεις στην νομοθεσία και το περιορισμένο πεδίο εφαρμογής. Αυτό είναι κάτι το οποίο εξετάσαμε πολύ σοβαρά στο πλαίσιο της πράξης προσβασιμότητας και είναι απαραίτητο να τεθούν τα, αυτά τα θέματα επιτάπητος ώστε κατά τη συζήτηση της νομοθεσία αυτής να είμαστε φιλόδοξοι και να έχουμε περιορισμένο αριθμό παρεκκλήσεων ώστε πράγματι να πρόκειται για παρεκκλήσεις και όχι για το σύνηθες. Αυτό λοιπόν είχαμε κατά νου και κατά την εκπόνηση της πράξης για την προσβασιμότητα, ε, γνωρίζοντας και αυτές τις εμπειρίες. Έτσι λοιπόν ε, έχουμε πληροφορίες σχετικά με τα τερματικά αυτοεξυπηρέτησης και την παροχή πληροφοριών. Ήθελα απλά να προσθέσω αυτά σε αυτά που είπε η συνάδελφο. Σας ευχαριστώ. Είναι ασυνήθιστο και πολύ ικανοποιητικό ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να είναι ακτιβίστρια, όχι μόνο γραφειοκρατική λειτουργία. Ο κύριος, ε, η συνάδελφος τώρα και μετά ο κύριος Μαριάς. Ευχαριστώ, ήταν θαυμάσιο αυτό το οποίο ακούσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τρομερό ενδιαφέρον η αναφορά την οποία μας παρουσίασε η Ρωμίνα. Η Ρουμανία έχει επικυρώσει την σύμβαση των, των Ηνωμένων Εθνών, ίσως να είναι και η τελευταία χώρα όμως η οποία δεν έχει επικυρώσει τις εφαρμοστικές πράξεις. Είναι προφανές ότι η πρόσβαση στις μεταφορές είναι απαραίτητη για να υπάρξει ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων με αναπηρίες. Αυτοί με την, οι άνθρωποι με περιορισμένη κινητικότητα απαιτούν να έχουν τις κατάλληλες συνθήκες έτσι ώστε να μπορούν να ταξιδεύουν όπως και όλοι οι υπόλοιποι πολίτες. και πράγματι η διαδικασία αυτή προειδοποίησης ε, ε, είναι πράγματι πάρα πολύ ε, επώδυνη η διαδικασία αυτή. Επίσης και οι διαδικασίες οι οποίες ισχύουν για τα ταξίδια μακράς διάρκειας, οι συνθήκες αυτές είναι απαράδεκτες και ουσιαστικά όλα τα άρθρα ε, της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών και ε, η Σύμβαση, η χάρτας ε, μάλλον των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν γίνονται σεβαστές. Στην ουσία αποφάσισαν αυτό το οποίο εθελοντικά μπορούν να εφαρμόσουν για μία πενταετία αρνούνται να το εφαρμόσουν, δεν εξυπηρετούν τους ταξιδιώτες, ε, επιβάτες ε, με αναπηρίες και το θέμα είναι να κατανοήσουν ότι μια κυβέρνηση δεν είναι απλά εκεί για να εφαρμόζει μόνο τις ρήτρες τις υποχρεωτικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά το σύνολο των προβλέψεων που ισχύουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και το επιχείρημα το οικονομικό δεν έχει εδώ καμία ισχύ γιατί είναι η απόλυτη προτεραιότητα η κάλυψη των αναγκών των ανθρώπων αυτών. Λοιπόν, θα συμφωνήσει και ο Έλληνας συνάδελφος με αυτά τα οποία λέω. Είναι ιδιαίτερα δραστήριος και αυτό σε σχέση με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα μπορούσαμε να οργανώσουμε μια επίσκεψη επιτόπου στην Ρουμανία και να μπορέσουμε να πιέσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Γιατί οι αποφάσεις οι δικές μας σαν Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν είναι δεσμευτικές φυσικά. Αλλά παρόλα αυτά όταν πηγαίνουμε σε μια χώρα προκαλούμε τις συνειδήσεις, αναγκάζουμε τους ανθρώπους να δουν με διαφορετικό τρόπο τα πράγματα και να κινητοποιηθούν αλλάζοντας μερικές φορές τις απόψεις τους. Και το θέμα δεν είναι μόνο οι μεταφορές ε, με τον σιδηρόδρομο αλλά ε, και σε άλλα θέματα της καθημερινότητας αντιμετωπίζουν δυσκολίες οι άνθρωποι αυτοί σε χώρες όπως η Ρωμανία. Και στον τομέα της εκπαίδευσης θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ανοίξουμε ε, τους, τις πόρτες αυτών τους ανθρώπους να μπουν στην αγορά εργασίας. Έχουν δικαίωμα οι άνθρωποι αυτοί να ενταχθούν και στην αγορά εργασίας και δεν θα πρέπει οι θέσεις αυτές εργασίας να είναι προστατευόμενες θέσεις ε, χωρίς καμία αξιοπρέπεια. Θα πρέπει να είναι θέσεις οι οποίες να είναι άξιες του επίπεδου των ανθρώπων αυτών και ε, χρήσιμες και για το πρόσωπο το συγκεκριμένο αλλά και για την επιχείρηση ή την υπηρεσία που τον απασχολεί. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θα ήθελα να προτείνω μία επίσκεψη λοιπόν στην χώρα σας να έρθουμε σε επαφή με τις αρχές έτσι ώστε να μιλήσουμε όχι μόνο για το θέμα των μεταφορών αλλά γενικότερα για τη θέση των ανθρώπων με περιορισμένη κινητικότητα στο σύνολο της ζωής στη Ρουμανία. Ο κύριος Μαριάς. Καταρχάς, ε, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ την αναφέρουσα για την ε, ανάλυση που μας έκανε και για την πρωτοβουλία της να φέρει την υπόθεσή της εδώ στην Επιτροπή μας αποδεικνύεται δυστυχώς ότι τα πράγματα στη Ρουμανία είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα για τα άτομα με αναπηρία. Ε, και από ό,τι φαίνεται οι αρχές δεν δείχνουν και ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μάλλον αξιοποιούν διάφορα παραθυράκια νομικά που υπάρχουν, ούτω ώστε να μην ε, ρυθμίσουν έτσι τα ζητήματα, ούτω ώστε να υπάρχει προσβασιμότητα. Ε, το γεγονός ότι μας είπε η αναφέρουσα ότι πρέπει προ 15 ημερών να ειδοποιήσει ότι πρόκειται να κάνει ένα ταξίδι και αν θα της δώσουν άδεια ότι δεν υπάρχει πρόσβαση στο σιδηρόδρομο, ότι δεν μπορεί να φτάσει μέχρι το σιδηροδρομικό σταθμό, ότι δεν μπορεί να ανέβει στο, στο τρένο. Αυτά τα πράγματα ε, κυριολεκτικά είναι, είναι απαράδεκτα. Ε, το θέμα είναι πώς μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε πρακτικά για να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Ε, πρώτα απ' όλα συμφωνώ με την ε, συνάδελφο, την Αστάρας, ε, που είπε ότι θα μπορούσε να γίνει μια επίσκεψη στη Ρουμανία. Και συζητώντας χθε για τις επισκέψεις, ουσιαστικά καταλήξαμε μόνο σε μια επίσκεψη και έχουμε αφήσει ανοιχτό το θέμα μιας επίσκεψης σε ένα άλλο κράτος πέλος. Νομίζω ότι αυτή η υπόθεση στην Ρουμανία ε, πραγματικά αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι αφορά χιλιάδες συμπολίτες μας και κυρίως αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι μάλλον η αναλγησία των αρχών των ρουμανικών που δεν ενδιαφέρονται να πάρουν συγκεκριμένα μέτρα. Έχω και μια δεύτερη πρόταση για να μπορέσουμε να ασκήσουμε όσο μπορούμε μεγαλύτερη πίεση διότι με βάση αυτά που είπε η Επιτροπή η οποία πραγματικά ενεργεί ε, με ένα ακτιβιστικό τρόπο υπέρ των ε, ατόμων με αναπηρία αλλά από ό,τι μας είπε υπάρχουν εξαιρέσεις, θα έρθει ένας νέος κανονισμός μέχρι να ψηφιστεί ο νέος κανονισμός θα περάσουν δύο χρονιά και οι φίλοι μας από τη Ρουμανία δεν θα μπορεί να μετακινηθεί. Λέω λοιπόν ως πρόταση να στείλουμε την ε, αναφορά της πρώτα απ' όλα στην Επιτροπή Μεταφορών και δεύτερον στην Επιτροπή Προϋπολογισμού και να ζητήσουμε από τους συναδέλφους να μην εγκρίνουν κονδύλια για τη Ρουμανία στο πλαίσιο των κονδυλίων που παίρνει και παίρνει αρκετά κονδύλια για τις μεταφορές και για άλλα θέματα μέχρι ότου να δώσει τα πρώτα δείγματα γραφής ότι ξεκινάει τη διαδικασία συμμόρφωσης. Αν λοιπόν από εδώ ένα μεγάλο μέρος των κονδυλίων, γιατί εμείς εγκρίνουμε τα κονδύλια ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αν λοιπόν αναστείλουμε ορισμένα κονδύλια για τη Ρουμανία, τα οποία είναι αρκετά εκατομμύρια, ίσως και δισεκατομμύρια, να είστε βέβαιοι ότι η ρουμανική κυβέρνηση θα έρθει πολύ γρήγορα να μας εξηγεί πώς πρόλαβε να ρυθμίσει όλα τα θέματα για την προσβασιμότητα στους σιδηροδρομικούς σταθμούς. Επειδή λοιπόν πιστεύω ότι η επίσκεψη θα συμβάλλει πράγματι για να ευαισθητοποιήσει την κατάσταση, αλλά επειδή πιστεύω ταυτόχρονα να περάσουν χρόνια μέχρι να αναγκαστούν οι ρουμανικές αρχές να ακολουθήσουν τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουν από τις διεθνείς συμβάσεις, εάν λοιπόν ε, θέσουμε το θέμα ε, στην Επιτροπή Μεταφορών και στην Επιτροπή Προϋπολογισμού αλλά και στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εγώ τουλάχιστον εκεί είμαι μέλος. Να αρχίσουμε λοιπόν να ασκήσουμε μια πίεση. Να σταματήσουμε να δίνουμε κονδύλια στη Ρουμανία. Τότε θα δείτε ότι θα συμμορφωθεί η κυβέρνηση της Ρουμανίας. Και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το πάρουμε έτσι ζεστά το θέμα, γιατί αλλιώς θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια μέχρι ότου να συμμορφωθεί η Ρουμανία και φυσικά οι φίλοι μας ε, και όσοι άλλοι έχουν προβλήματα κινητικότητας, αναπηρίας θα μείνουν εκτός εργασίας, δεν θα μπορούν να πάνε ε, για σπουδές, δεν θα μπορούν να μετακινηθούν και θα έχουν αυτές τις απαράδεκτες ε, συνθήκες. Και νομίζω ότι όσο δύσκολο και αν είναι αυτό και για τους συναδέλφους από τη Ρουμανία θα πρέπει επιτάπητος να τεθεί διότι φοβάμαι ότι θα περάσουν πολλά χρόνια για να συμμορφωθεί η ρωμανική κυβέρνηση. Αν πάρουμε αυτά τα μέτρα ίσως καταφέρουμε κάτι σημαντικό για τους συμπολίτε μας που είναι στη Ρουμανία. Ευχαριστώ. Thank you very much. Would you like to take... Ευχαριστώ πολύ. Θέλετε ξανά τον λόγο. Για να είμαι ειλικρινής, είναι εξαιρετικό να βλέπω τόσο μεγάλη στήριξη για το σκοπό αυτό. Συμφωνώ ότι πρέπει να γίνει κάτι. Ε, οι κατευθυντήριες γραμμές σίγουρα δεν έχουν αποτέλεσμα για τη ρουμανική κυβέρνηση. Τους έχουν δοθεί τόσες υποχρεώσεις που αν μπορέσουν να το παρακάμψουν θα το παρακάμψουν και θα κάνουν ό,τι μπορούν. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει κάτι πιο δραστήριο όπως αυτό που προτείνεται. Νομίζω ότι έτσι μπορούν να διορθωθούν τα πράγματα. Αν περιμένουμε από τη ρουμανική κυβέρνηση να βελτιώσουν το σιδηροδρομικό του δίκτυο και να υπάρχει μεγαλύτερη πρόσβαση, μπορεί να μην φτάσω να το δω εγώ πριν από τη σύνταξή μου. Ε, χρειάζεται κάτι πιο δραστήριο, κάτι που θα τους κινητοποιήσει. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ που ταξιδέψατε μέχρι εδώ για να μοιραστείτε μαζί μας την ιστορία σας. Η αναφορά είναι πάρα πολύ σημαντική, προφανώς και θα μείνει ανοιχτή, προφανώς και θα την στείλουμε και στην Επιτροπή Μεταφορών για γνωμοδότηση εν ώψη της ε, ε, έκθεσης για την ε, εφαρμογή των σιδηροδρομικών δικτύων είναι πάρα πολύ σημαντική επιρρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι λοιπόν ένα καλό παράθυρο ευκαιρίας να αναλάβουμε δράση και πρέπει και εμείς εδώ στην Επιτροπή μας να ε, κινητοποιήσουμε τα μέλη που έχουμε. Υπάρχει ένας ε, ο οποίος είναι πληρωτής στην Επιτροπή Μεταφορών, η Ρώσα και έχουμε και άλλους στην Επιτροπή Επιτροπή Αναφορών που είναι είτε τακτικά είτε αναπληρωματικά μέλη στην Επιτροπή Μεταφορών και θα τους ζητήσουμε να παρακολουθήσουν προσεκτικά το ζήτημα ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι θα μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Άλλωστε η ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων τι είναι αν δεν περιλαμβάνει και τα άτομα με αναπηρία και αναφερόμαστε σε ελεύθερη κυκλοφορία από τη μία χώρα στην άλλη για σκοπούς εργασίας, σπουδών ε, και οικογένειας. Το να μπορεί κάποιος ε, να κινηθεί και εντό της χώρας του με τα βασικά μεταφορικά μέσα, τι σημαίνει ελεύθερη κυκλοφορία αν δεν μπορεί να το κάνει. Ε, αν είναι απλώς όνειρο απατηλό για κάποιους ανθρώπους ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα και το να πάρει ένα ε, μέσο μαζικής μεταφοράς στη χώρα του. Είναι πραγματικά εφιάλτης αυτό και πραγματικά πιστεύω ότι είναι πονίδιστο το γεγονός ότι οι ρωμανικές αρχές ε, καταχρώνται τις εξαιρέσεις στην νομοθεσία και όπως είπε και ο κύριος Μαριάς τις χρησιμοποιούν ως παραθυράκι για να μην συμμορφούνται. Ε, δεν είναι σίγουρα καλό κάτι τέτοιο. Θα στείλουμε λοιπόν μια πολύ αυστηρή επιστολή στις ρωμανικές Αρχές ε, και να ζητήσουμε την άποψή τους για το θέμα, ιδίως ε, ε, για τις εξαιρέσεις που τους δόθηκαν στον κανονισμό, κάτι το οποίο δεν θα συνεχίσει να ισχύει διαπαντός, επομένως πρέπει να κάνουν κάτι γι' αυτό. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνουμε και από εκεί και πέρα φυσικά θα το ε, παραπέμψουμε και στη γραμματεία για την επόμενη φορά που συζητήσουμε σχετικές διερευνητικές αποστολές να δούμε αν μπορούμε να κινητοποιήσουμε συναδέλφους και πολιτικές ομάδες για να ε, υλοποιηθεί η αποστολή. Όσον αφορά την Επιτροπή Προπολογισμών, τη σχετική αναθεώρηση και την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού, ε, δεν ε, είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής να κάνει τίποτα από αυτού, αλλά βασιζόμαστε στα μέλη της Επιτροπής που είναι και μέλη στις ε, Επιτροπές αυτές για να τα εξετάσουν. Ιδίω εσείς κύριε Μαριά. Προσέξτε το λοιπόν το θέμα. Και τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι οι διεθνείς υποχρεώσεις ε, για τις οποίες έχει δεσμευθεί η Ρουμανία όταν ακυρώσουν τη σύμβαση θα ε, αρχίσουν να ισχύουν και θα φροντίσουμε να τους ενημερώσουμε γι' αυτό για άλλη μια φορά με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ σε όλους για αυτή την πρωινή συνεδρίαση. Καλή όρεξη σε όλους και για σας που ήρθατε από την ε, Ρουμανία τις καλύτερες ευχές μας στους φίλους σας και τους υποστηρικτές σας και να συνεχίσετε τον αγώνα.